So, ladies and gentlemen, dear colleagues, please take a seat. Good. dann kommen wir zu Punkt 2. Περνάμε στο σημείο λοιπόν 2 τη ημερήσιας διάταξη, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αιτήματα για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξη, αν όχι την εγκρίνουμε ω έχει. Υπό το σημείο 3 έχουμε την έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίασης της 9 η Νοεμβρίου. Εάν λοιπόν εάν, ε, δεν ε, υποβληθούν αιτήματα για τροποποίηση των πρακτικών αυτών ω το τέλος της σημερινής συνεδρίας, θα θεωρούσουμε πώ έχουν εγκριθεί. Περνάμε στο σημείο 4 τώρα. εδώ από τη Λισαβόνα ως το Λούνεμπορκ και από το Ταλίν έως την Ταμίνα. Καλωσορίζω όλου όλους μας τους τηλεθεατές μέσω web streaming. Μας παρακολουθούν από τις οθόνες τους αφού έχουμε web streaming στη σημερινή μα συνεδρίαση και γι' αυτό βέβαια σας καλώ όλους να μιλάτε αργά και καθαρά έτσι ώστε να ακούγεται σωστά και η διαρμηνία. και βέβαια να φέρεστε με τρόπο τέτοιο που να πείθετε τους τηλεθεατές μας ως προς τις εργασίες που κάνουμε εδώ. Ε, τώρα, έχω μια ιδιαίτερη ανακοίνωση. Ε, δίπλα από τον Μάρτιν κάθεται ο Λέων, ο οποίος ε, μας είναι γνωστός, γιατί εδώ και 7 χρόνια εργάστηκε στη γραμματεία της Επιτροπής μας και παρακολούθησε μια σειρά από σημαντικούς φακέλους της Επιτροπής μας και έχουμε εκτιμήσει πάρα πολύ την ήρεμη συμπεριφορά του, όχι πάντοτε βέβαια. Και δυστυχώς θα χρειαστεί ο Λεό να μας εγκαταλείψει λόγω των απαιτήσεων κινητικότητας του προσωπικού. καθώς ε, θα μεταφερθεί στην ε, μονάδα για τις δεταλικές ε, σχέσεις και το G8. Δηλαδή θα αρχίσει να ασχολείται πλέον με ε, ζητήματα ακόμα υψηλότερου πολιτικού επίπεδου. Είμαστε πολύ λοιπόν, Λέων, που μαθαίνουμε στις εγκαταλείψεις. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο πλαίσιο των ε, περαιτέρω εργασιών και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Ε, ε, Λέων. Ελπίζω να είσαι εδώ στις 6.30 γιατί θα έχουμε ένα μικρό ποτό χριστουγεννιάτικο στο εστιαστόριο στο Ιένα. Στο μεσογειακό εστιατόριο όπως λέγεται, δηλαδή πρέπει να πάει κανεί στο 0, στο ισόγειο, μετά να περπατήσει ολοκύτω διάδρομο για να φτάσει στο Ιένα, οπότε ελπίζω να σας δω όλους εκεί για αυτό το Christmas drink. έτσι ώστε να συζητήσουμε λίγο και τα όσα μας απασχόλησαν φέτος. Περνάω λοιπόν τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την πρώτη μας ψηφοφορία για σήμερα. Ως συνήθως θεωρώ ότι έχετε όλοι τις κάρτες σας για την ψηφοφορία, οπότε ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Οπότε βλέπουμε πως λειτουργήσε καλά. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5 και στην κανονική πλέον ψηφοφορία, την πραγματική ψηφοφορία, η οποία έχει να κάνει με τις εκτελεστικές αμμοδιότητες, τα implementing powers. Πρώτη λοιπόν τροπολογία, υπαριθμό 14 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Block vote. Μαζί δηλαδή με την 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά στην ελέγξουμε τη 15. Άρχεται λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άρα σημαίνει σε σχέση με τον blog του δεν περάσε. Περνάμε λοιπόν στο πλογιά 16. Δώστε μου μισό λεπτό, Πρόεδρος. 18 περνάμε. Στην τροπολογία 18. Σε δύο τμήματα. 18 λοιπόν πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν το πρώτο τμήμα της 18, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 18. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5. Και την 3 μαζί με αυτήν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. περνάμε στην τροπολογία 19. Με προφορική τροποποίηση oral amendment υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για να είμαστε λίγο προσεκτικοί τώρα εδώ. Απολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 την εξετάσαμε. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία επί του συνόλου του εγγράφου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία Και εγκρίνεται λοιπόν με μεγάλη πλειοψηφία. Θα θυμάμαι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης προφορικό ερώτημα σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο για, την, ε, για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες. Μία και μόνη ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Και σχεδόν ομόφωνα εγκρίνεται και αυτή η προφορική ερώτηση. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις προφορίες μας για σήμερα. Περνάμε στο σημείο 7 της μερίσιας διάταξη. Η ερμηνεία και υλοποίηση ε, της Διοργανικής Συμφωνίας. Όπως ε, γνωρίζετε στι 13 Απριλίου του 2016 αποφασίστηκε αυτή η Διοργανική Συμφωνία η οποία περιλαμβάνει πολλά καινοτόμα στοιχεία και έχει και βέβαια και μια σειρά από πολιτικού χαρακτήρα επιπτώσεις ε, και προτού δώσω το λόγο στον εισηγητή μας θα ήθελα να σας πω ότι ένα τμήμα αυτής της διοργανική συμφωνίας ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί σε ό,τι αφορά δηλαδή τις εξωτερικές διαστάσεις και σε ό,τι αφορά αυτό το τμήμα της διοργανικής συμφωνίας βρισκόμαστε ε, σε διαπραγμάτευση εδώ και 1,5 χρόνο με τις διάφορες προεδρίες του Συμβουλίου. Αλλά μέχρι στιγμής το Συμβούλιο δεν κατάφερε να αποδεχτεί τα δικαιώματα εκείνα τα οποία έχουν κατοχυρωθεί για μας για το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Δηλαδή, συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ε, πληροφορίες ε, οι οποίες αφορούν το σύνολο του κύκλου ζωής εντός εισαγωγικών μιας συμφωνίας, δηλαδή από την εντολή διαπραγμάτευσης ε, που δίνεται έως τα επιμέρους τμήματά της και σε ό,τι αφορά και την εφαρμογή της στην πράξη. Και από εκεί και μετά αυτή η αυτόματη και άμεση διαβίβαση των εντολών ως δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει και αυτή απορριφθεί από το Συμβούλιο, όπως επίσης και η αξίωσή μα να μην είναι δυνατή η προσωρινή εφαρμογή μια τέτοια συμφωνία εάν δεν έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από εκκρεμή στοιχεία επί των οποίων διαπραγματευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο αλλά για τα οποία το Συμβούλιο δεν κατάφερε να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του πράγμα βέβαια το οποίο είναι λυπηρό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δική μας διαπραγματευτική ομάδα να εξετάζει το εάν θα είχε νόημα να προσφύγουμε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν το Συμβούλιο δεν προβεί σε κάποιες παραχωρήσεις στο πλαίσιο της διαπραγματεύσής μας. Ε, ένα στοιχείο το οποίο με εκνεύρισε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά δικότερα την πρόσβαση στις διάφορες εντολές είναι το εξή. Ε, ζητήσαμε την εντολή τη διαπραγματευτική σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση με το Μαρόκο πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης καν στο πλαίσιο δηλαδή της, ε, των όσων προβλέπει η συνθήκη. Αλλά λάβαμε μια επιστολή που μας έλεγε τι, ότι βρισκόμαστε ακόμα σε διαπραγμάτευση και αν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο μηχανισμό θα εφαρμόζουμε, δεν μπορούμε να σα διαβιβάσουμε αυτή την εντολή. Κάτι τέτοιο είναι πραγματικά θράσος από την πλευρά τους να τοποθετήσουμε αυτόν τον τρόπο απέναντί μας. Άρα λοιπόν αυτό το τμήμα της Διοργανικής Συμφωνίας παραμένει σε κρεμότητα. Ωστόσο το υπόλοιπο ε, ήδη ισχύει, ήδη εφαρμόζεται και ο Μπέντσεν θα μας ενημερώσει σχετικά κάνοντας μια εισαγωγική παρέμβαση. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Θα γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πρόκειται να συνάψουμε μια νέα θεσμική συμφωνία προκειμένου να βελτιωθούν οι λειτουργίε μεταξύ των θεσμών το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας εδώ γίνεται στην ΑΦΚΟ και στη ΙΟΕ. Αλλά υπάρχουν θέματα που άπτονται διεθνώ συμφωνιών και το Κοινοβούλιο εκεί έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Και είναι σημαντικές οι σχέσεις να είναι καλές. Αν θέλουμε να αναλάβουμε σοβαρά αυτή την ευθύνη. Έχω δύο προβληματισμούς. Η προσωρινή εφαρμογή. Η ιδιαίτερη προτεραιότητα για μένα είναι όταν θεωρείται δεδομένη η συνένεση του Κοινοβουλίου. Αναφέρεται στις ε, συμφωνίες ο διαχωρισμός των εξουσιών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει τη σύμφωνη γνώμη στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ή αποφασίσει να αρνηθεί και αυτό καθιστά κενό περιεχομένου και περιεχομένου τη συμφωνία. Αυτό το δικαίωμα είναι κάτι που είναι βασικό δικαίωμα της συνθήκης και η Πολιτική Επιτροπή, το Συμβούλιο θα πρέπει να σεβαστεί. Δυστυχώς Έχουμε δει αρκετά παραδείγματα που προσπάθησε αυτό να το βάλει στην άκρη η Επιτροπή. Κάτι που δεν είναι προσωρινό από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για το πότε αρχίζει να εφαρμόζεται. Και αυτό συνέβη πριν από 1,5 χρόνο όταν η Επιτροπή έκανε μια συμφωνία με την Νορβηγία. Αυτό το κοινοβούλιο έχει άποψη σχετικά με την απόφαση του, της Νορβηγίας για τους δασμούς. Το 2013 ζητήσαμε από την ΕΠΗ να αναλάβει δράση. Η Επιτροπή φαίνεται να γνώρισε τις απόψεις του Κοινοβουλίου και έκανε μια συμφωνία με την Νορβηγία. Για να χειροτερέψουν τα πράγματα, η Επιτροπή αποφάσισε να υπάρξει προσωρινή εφαρμογή και συνεπώς η απόφαση ήταν άσχετη. Αυτό πραγματικά είναι μία ντροπή και νομίζω ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά. Από ό,τι φαίνεται όμως το Συμβούλιο και η Επιτροπή Εξωτερικών Υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να παίρνουν αυτά στα σοβαρά σε ό,τι αφορά την εντολή διαπραγμάτευσης. Όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες, αλλά η τελική εντολή είναι άμεσα προσβάσιμη. Σύμφωνα με το άρθρο 2008 το, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερωθεί σε όλες τις φάσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα με τρίτες χώρες. Σε ό,τι θα πρέπει αυτά να τα μοιραστούμε με το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να τον, το τονίσουμε. Θα ήθελα να δω τι έχουν να πούν και οι άλλες ομάδες. Thanks a lot. Who wants to take the floor? Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, Έμα, παρακαλώ. Thank you. Um, the ECR group views the improvement of our Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Θέλουμε και, θεωρούμε και εμείς ότι πρόκειται ε, αυτή η προσπάθεια είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει και την ανταγωνιστικότητά μα αλλά και θα προωθήσει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τις, ε, την πρόοδο που έχει σε αυτό το επίπεδο η Επιτροπή μαζί μα. Και επίση συγχαίρουμε την Επιτροπή ε, για τι προσπάθειε που έχει κάνει σε ό,τι αφορά την αύξηση τη διαφάνεια ε, και την συνεχή επαφή με τη δική μα Επιτροπή. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη βελτιωμένη συνεργασία, αυτή τη ε, βελτιωμένη ατμόσφαιρα, θα θέλαμε να δούμε μια αντίστοιχη προσπάθεια και από την πλευρά του Συμβουλίου. Δηλαδή, ε, καλύτερο συντονισμό σε ό,τι αφορά την νομοθετική διαδικασία, σε ό,τι αφορά δηλαδή καλύτερα χρονοδιαγράμματα, αλλά και καλύτερη εξέταση των νομοθετικών προτάσεων, στο πλαίσιο δηλαδή των όσο προβλέπει και το άρθρο 35 τη Συμφωνία, αλλά και η οθέτηση των σχετικών συστάσεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Επίση, θα, πρέπει, θα πρέπει οι κατευθυντήρε γραμμέ διαπραγμάτευση από την πλευρά του Συμβουλίου να έρχονται τώρα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνεχή διαβούλευση και με όλου του συναρμόδιου φορεί σε όλε τι φάσει τη διαπραγματευτική διαδικασία τέτοιου είδου συμφωνιών από, από την αρχή Τη ε, όλη διαδικασία έτσι ώστε να αποφύγουμε καταστάσει όπω αυτή τη ΣΥΤΑ δηλαδή στο παραπέντε των εισαγωγικών. Και επίση είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει αξιολογήσει αντικτύπου έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, τέτοιου είδου αξιολογήσει θα πρέπει να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τι ανάγκε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, δηλαδή η ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αποτελεί ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία είναι ενδυμικά σε κάποια κράτη-μέλη αλλά όχι σε άλλα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν στόχοι οι οποίοι είναι ενιαίοι και οι οποίοι ε, προσπαθούν να αποφύγουν, αν θέλετε, να προλάβουν ένα σωρευτικό άχθος σε τέτοιου είδους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, και επίσης θα πρέπει μέσω της ε, εμπορικής μας πολιτικής να έχουμε πάντοτε κατά νου συγκεκριμένα οράματα σε αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς παραμένουμε, εμένουμε στα Στι αρχέ, τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα, και κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλαμβάνει δράση εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται και όχι όπου είναι περιττή η δική τη παρέμβαση. Ευχαριστούμε, Χέλμουτ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εμφαντικά τον εισηγητή για αυτή την σύντομη εισαγωγή που έκανε. Θεωρούμε και εμείς πως η καλύτερη νομοπαραγωγή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, ειδικότερα εάν το εξετάσουμε ακριβώς υπό το φως της σύναψης νέων εμπορικών συμφωνιών. Σε δύο στοιχεία θα ήθελα να αναφερθώ, ε, τα οποία ε, δείχνουν να είναι ιδιαίτερα επίκαιρα και έχουν τεθεί ε, εκ νέου προς παρότι θεωρούσαμε πως είχαν ολοκληρωθεί. Πρώτο λοιπόν είναι η διαφάνεια ε, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαπραγμάτευση και από την πλευρά όλων των μερών. Και αυτό είναι το εξή. Όταν ε, το Συμβούλιο ζητάει από την Επιτροπή να επεξεργαστεί μία εντολή και εμεί ε, καλούμαστε να συντάξουμε ένα ψήφισμα από την πλευρά μα για οποιοδήποτε ζήτημα, γιατί εντάξει μπορεί να αφορά το διεθνέ εμπόριο αλλά μπορεί να αφορά και άλλες επιτροπέ που σχετίζονται με ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, ήδη στο πλαίσιο δηλαδή του συντονισμού που θα γίνεται μεταξύ Συμβουλίου επιτροπή και Κοινοβουλίου, θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια. Δεν μπορεί δηλαδή στο πλαίσιο τη διαπραγμάτευσης με τη Μερκοσούρ να υπάρχει λιγότερη διαφάνεια σε σχέση με τα όσα είχαμε στο πλαίσιο της TTIP, σε σχέση με τα όσα είχαμε επιτύχει στο πλαίσιο της ΕΝΤΑ ε, στο πλαίσιο προσπαθήσαμε εκεί δηλαδή να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και ούτω καθεξής. Ό,τι έχει τύχει διαπραγμάτευση μέχρι τώρα ουσιαστικά δεν ήταν πλήρω προσβάσιμο σε εμά. Πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Άρα λοιπόν, εκείνο που θα πρέπει να μα απασχολήσει είναι το πώ θα μπορέσουμε στην ίδια την νομοθεσία, απριόρι εκ των προτέρων, να υπάρχει μια τέτοια βελτίωση της διαφάνειας στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων. Το δεύτερο τώρα στοιχείο, η δεύτερη διάσταση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ είναι το εάν ή όταν έχουμε διαβουλεύσεις με τους διάφορους συναρμόδιους φορείς, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τις επιχειρήσεις, τότε κατά κανόνα ο επιχειρηματικός κλάδος πάντοτε συμμετέχει. Ε, πράγμα το οποίο είναι λογικό, αλλά συχνά δεν συμμετέχει η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο τη νομοθεσία και πάλι θα πρέπει να εξετάσουμε το πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε δομέ και μηχανισμού οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη και ε, τα συμφέροντα που εκπροσωπεί, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και τελικά και το ίδιο το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να αξιώνουμε να αξιώσουμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος στο πλαίσιο της επικοινωνίας που θα έχουμε με την Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη και αυτές τις διαστάσεις, αυτές τις τοποθετήσεις, αυτές τις οπτικές γωνίες, ειδικότερα ακριβώ και στο πλαίσιο της ε, εντύπωση ε, που έχει η κοινή γνώμη, στο πλαίσιο αυτών των ε, συμφωνιών, αλλά και των συμφωνιών, για παράδειγμα, διασύνδεσης. Στο πλαίσιο λοιπόν εδώ της βελτίωσης της νομοθεσίας θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά εάν θέλουμε η πολιτική ε, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά προς το συμφέρον των πολιτών μας. Ευχαριστώ, Λεωπρόεδρο Αλήση. Ε, Έχω πολύ λίγα να προσθέσω στα όσα είπε και ο συγητής και οι συνάδελφοι, γιατί μας βρίσκουν σύμφωνος πολλά από τα σημεία που ετέθησαν. Η ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών πάντοτε τόνισε ότι θα έπρεπε να γίνουν βήματα μπροστά σε επίπεδο διαφάνειας. Ορισμένα βήματα έγιναν από την Επιτροπή, αλλά με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αντίσταση του Συμβουλίου ως προς την εφαρμογή διαδικασιών που συμπεριλαμβάνουν το Κοινοβούλιο σε όλες τις διαδικασίες πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επιμείνουμε σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο αλλά είναι σημαντικό να ασκήσει την ίδια πίεση και η Επιτροπή ως εγγυήτρια του νέου τρόπου αυτού εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων ξεκινώντα από το Κοινοβούλιο. Αν η Επιτροπή, δεν μπορεί να απουσιάσει από μία άμεση τέτοιου είδους δράση. Δεύτερο σημείο, Θεωρούμε, πέρα από όσα ήδη αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους, ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να εμπλακεί όχι μόνο στη βάση διαπραγμάτευσης των διαφόρων συμφωνιών, ξεκινώντας από τις πρώτες σελίδες, αλλά όλες τις φάσεις ελέγχου ήδη μπορέσαμε να συζητήσουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα της Επιτροπής να συμπεριληφθεί παρατηρούν σε, ε, σε όλες τις διαδικασίες το Κοινοβούλιο που θα μπορέσει να δράσει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ή μη εφαρμογή ορισμένων σημείων, κυρίως ε, λόγω του ότι κεφάλαια τα οποία ήταν υπολοιματικά, όπως αυτό για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τώρα αρχίζουν να αποκτούν ως όλο και πιο μεγάλο βάρος και, και ιδίως το θέμα της εφαρμογής και της εναρμόνισης των κανονισμών. Θεωρούμε λοιπόν ότι και σε ό,τι αφορά το σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε την ανάγκη ε, να ε, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια με το Κοινοβούλιο. Ε, Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Ιωάννα Λεσούκ, λοιπόν, από την Ευχαριστώ που καλέσατε την Επιτροπή να λάβει το λόγο, Πρόεδρε. Η διαθεσμική συμφωνία για βελτίωση του μελλοντικού έργου είναι σημαντική, διότι μας βοηθά να συνεργαζόμαστε καλύτερα, αλλά να καταλήγουμε και σε καλύτερα αποτελέσματα. Θα ήθελα παρόλα αυτά να τονίσω ότι στις συζητήσεις οποιαδήποτε εισιτής για την εφαρμογή της συμφωνίας θα πρέπει να γίνει σε τριμερές επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεσπίζεται και στο άρθρο 9 της συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις γίνεται βάσει του άρθρου 13. Οι τεχνικές συζητήσεις γίνονται τώρα, τεχνικό επίπεδο συζητήσεις και τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτό ξέρουμε ότι είναι αν δεν καταλήξουν δύσκολο να συζητηθούν για τα πώς θα γίνονται όλες αυτές οι διεθνείς διαπραγματεύσεις. Στις 12 Δεκεμβρίου, όπως ξέρετε, θα υπάρξει μία συνεδρίαση πολιτικού περιεχομένου για να δούμε που ακριβώς βρισκόμαστε στο Στρασβούργο και εμείς θα αναλάβουμε τις διαθεσμικές μας ε, ε, δεσμεύσεις για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, σε αυτό το επίπεδο στα τρία θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Αυτό μπορώ να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σύμφωνος ότι έχουμε καταλήξει σε μία συμφωνία για τις 12 Δεκεμβρίου για να δούμε από πολιτική σκοπιά που βρισκόμαστε. Συμφωνήσαμε ότι ίσως την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε αυτή τη συνεδρία στην εβδομάδα του 12, της, 12, της 18ης Δεκεμβρίου, όχι της 12ης, δεύτερον, όσον αφορά το περιεχόμενο. Βεβαίως εδώ έχουμε στην Επιτροπή μας μια πολύ καλή πρακτική. Πιστεύω λοιπόν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζει στις διαπραγματεύσεις αυτή την πρακτική. Η σαφής μας άποψη είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία συμφωνία πριν εμείς να γνωμοδοτήσουμε, να συνενέσουμε ως κοινοβούλιο. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε αυτό το επίπεδο να καταλήξουμε όλες οι επιτροπές και όλο το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να είμαι σύντομος, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση και να πω ότι θα λάβω υπόψη όλα τα σχόλια στην επόμενη εκδοχή της έκθεσης που θα σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Βεβαίως, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις πως είπατε, σήμερα υπάρχει τεχνικού επίπεδου συνεδρίαση και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια κάποια βελτίωση του άλλου συστήματος μετά τη συνεδρίαση αυτή. Λοιπόν, θα συζητήσουμε στις 22 ε, Ιανουαρίου το σχέδιο έκθεσης, 26 Ιανουαρίου λίγη η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 20 Φεβρουαρίου συζήτηση στην Επιτροπή σας ευχαριστώ ολοκληρώνεται η συζήτηση του σημείου 7 περνούμε στο 8 θα ήθελα να καλέσω τον υπεύθυνο Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σιγκαπούρης να έλθει, να καθίσει στο βήμα δίπλα. την ε, ε, Υπουργό, με συγχωρείτε. So, item 8 is uh, the... Uh, λοιπόν είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ε, συμφωνία ε, με την Σιγκαπούρη για το ελεύθερο εμπόριο. Έχει συζητηθεί αυτό το θέμα ήδη. Η... Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χρειάστηκε να απαντήσει πολλές ερωτήσεις της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως όσον αφορά ποια είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι από κοινή. Στις 16 Μαΐου δημοσιεύτηκε η απόφαση αυτού του θέματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τώρα γνωρίζουμε ποιε είναι μέσα αφήνεια, ποιε είναι οι αποκλειστικέ αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκή είναι οι από κοινού ε, αρμοδιότητες. Υπάρχουν δύο ε, στοιχεία που αφορά τις επενδύσεις και την διευθέτηση των διαφορών στα οποία υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα στην συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό. Ότι θα πρέπει να υπάρχει στην συμφωνία κάποιο χωριστό κομμάτι. Εμείς ακολουθούμε αυτή την γραμμή σε τέτοιου είδους συμφωνίες όπου υπάρχουν τέτοιου είδους κοινέ εποκοινού αρμοδιότητες. Δηλαδή, ό,τι αφορά τις επενδύσεις για τη διαφορών. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταστήσαμε και απόλυτα σαφές στο ψήφισμα της ε, εντολής ε, για διαπραγμάτευση με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Έχει λοιπόν επιληθεί το θέμα αυτό, άρα μπορούμε να ασχοληθούμε περισσότερο με το περιεχόμενο της ε, συμφωνίας και για να το κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση υποδέχομαι δίπλα μου την υπεύθυνη Υπουργό Σιλάν από την Σιγκαπούρη σε θέματα εμπορίου και της δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Λάγκε για την ε, ευγενική εισαγωγή σας και σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε στα πλαίσια της ΦΙΤΙΕ e για, για σας. Όπως ε, ξέρουμε, παντού εμφανίζονται διάφορα προστατευτικά κινήματα, δεδομένου ότι υπάρχουν ε, σήμερα προβλήματα στο διεθνές Οι πιο ανεπτυγμένες ε, οικονομίες βλέπουν ότι διάφορες οι παραδοσιακές τους πολιτικές είναι κατά της παγκοσμιοποίησης και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης με τα πλαίσια των εμπορικών και βιομηχανικών πολιτικών. Η λύση δεν είναι να κλείσουμε τις αγορές, αλλά να μπορέσουμε να επωφεληθούμε δίκαια από τα ωφέλη της ε, παγκοσμιοποίησης. Εμείς είμαστε υπέρ του κράτους δικαίου, του ε, σεβασμού των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και θέλουμε να υπάρχει πολυμερή συνεργασία στα πλαίσια του εμπορίου. Θέλουμε να σεβαστούμε τους στόχους του ΠΟΕ για την εφόρο ανάπτυξη και να μπορέσουμε πάντα να σεβόμαστε διεθνείς συμφωνίες. Το εμπόριο είναι στο αίμα μας. Εμείς ε, πρέπει να πω ότι από τον 19ο αιώνα είμαστε στην Σιγκαπούρη ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Στη στρατηγική μας θέση στην, ε, στο μέσον μιας μεγάλης θαλασσίας οδού, πολύ σημασία, μας κάνει πάρα πολύ μεγάλο. Σήμερα είναι ε, ο όγκος του εμπορίου 3,5 φορές ανώτερος του ε, του ΑΕΠ μας και είναι ένας από τους λόγους της ευημερίας σας. Θέλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να ε, αναπτύξουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή τις 21 τέτοιου είδους ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με όλους τους παγκόσμιους συνεργάτες μας. Έχουμε υπογράψει τον Νοέμβριο την ε, συμφωνία με τις χώρες ΑΖΕΑΝ και περιμένουμε σύγχρονα την επικύρωση. Βεβαίως, ξέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι το TPP έχει αποχωρήσει ενζητέρους, η υπόλοιποι 11 έχουν μείνει και πιστεύουμε αυτό ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η Σιγκαπούρη επίσης θέλει να συνάψει και για μία ε, συμφωνία εμπορική με νέους εταίρους όπως την ε, Σρι Λάνκα και νέες ενός χωρών στην περιοχή μας. Ξέρουμε ότι το εμπόριο επίσης είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό εδώ και χρόνια και για σας ξέρουμε ότι η συνθήκη της Ρώμης βασίστηκε επίσης και στην εμπορική πολιτική και στην ευημερία και στο ελεύθερο εμπόριο. Σήμερα έχετε 38 εμπορικές συμφωνίες με 69 εταίρους και ξέρουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε και νέε φιλόδοξε συμφωνίε με τη Χιλή, με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία και άλλε χώρε. Στην παρούσα κατάσταση, λοιπόν, πρέπει να πω ότι είναι καθυσχαστικό το ότι ο πρόεδρο Γιούγκερ είπε, όταν μίλησε για την κατάσταση τη Ένωση, πόσο σημαντική είναι η πολιτική ελεύθερου εμπορίου. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερη εμπορική οικονομία ανά τον κόσμο. Είναι υπέρ της φιλελευθερωτής. Χαιρετίζουμε αυτή το νέο ε, ατζέντα για την απελευθέρωση του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σιγκαπούρη είναι ένας φυσικός εταίρος και αναλαμβάνει δεσμεύσει για την επιλογή. Δεν είναι τυχαίο το ότι είμαστε η πρώτη χώρα της ΑΣΕΑΝ με την οποία επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει διμερή συμφωνία FTA το 2009. Τη νέα αυτή συμφωνία είναι πολύ σημαντική διότι ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη συμφωνία. Πέραν λοιπόν της στρατηγικής της σημασίας πρέπει να πω ότι υπάρχουν ορατά και εφικτά κέρδη για όλες τις επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσουν οι επενδύσεις και το διμερές εμπόριο να αυξηθεί θα υπάρξουν εξαιτία, ε, χάρη στις παραδοσιακές ε, ε, συμφωνίες, προτιμησιακές συμφωνίες, άρση των εμποδίων και θα προστατευτούν όλα τα εμπορικά δικαιώματα. και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε και εκεί ότι η προώθηση των επενδύσεων θα πρέπει να ε, συμβαδίζει με την αηφόρο ανάπτυξη και να προστατεύσει τους λαούς. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έτσι, επειδή υπάρχει και ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ε, κοινωνική ευθύνη, για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ε, προστασία των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των φυσικών πόρων, πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Εμείς θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία διμερώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Σήμερα ε, είμαστε η τρίτος εμπορικός εταίρος και πιστεύουμε ότι επειδή είμαστε εσείς είστε οι τρίτος εμπορικός και εμείς είμαστε οι πρώτοι στην περιοχή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε λοιπόν για υπηρεσίες και εμπόριο η καλύτερο εταίρος πριν από την Ρωσία, την ε, ε, Ιαπωνία και υπάρχουν, έχουν ως έδρα τη Σιγκαπούρη περισσότερο από 13.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθώς και διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα και οργανώσεις οι οποίες εμπλουτίζουν τη ζωή. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να βελτιώσουμε τη σχέση μας, κυρίως το επόμενο χρόνο, δεδομένου ότι θα ε, ασκήσουμε την Προεδρία της ε, ΑΖΕΑΝ. Έτσι θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την ΑΖΕΑΝ ώστε να γίνει μια περιοχή ανθεκτική και με στόχο την ανάπτυξη. Με συνεκτικές πολιτικές πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε στα διάφορα οικονομικά μπλοκ, στις διάφορες αβεβαιότητες του εμπορίου και κυρίως θα μπορέσουμε να ε, ε, εστιάσουμε την προσοχή μας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην καινοτομία και σε άλλους σημαντικούς τομείς, στην ψηφιοποίηση του εμπορίου. Το 2016 αυξήθηκε 4,9 το ΑΕΠ του, ΑΣΕΑΝ και οι εξαγωγές είχαν ετήσια ανάπτυξη του 5,8% για κάποια χρόνια. Πρόκειται για μια εξαιρετικά μεγάλη αγορά που απευθύνεται σε πολλά εκατομμύρια ε, πολιτών. Είμαστε η ΑΣΕΑΝ είναι, όπως σας είπα, η τρίτος πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος. Και πρέπει να πω ότι έχει και πάρα πολλές συμφωνίες κλειδιά με άλλους ε, εταίρου στο εξωτερικό, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Κίνα και άλλες σημαντικές χώρες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η διμερής αυτής συμφωνία θα μας ευνοήσει όλους. Η FTA, η συμφωνία με την είπα πρέπει να πω ότι επίσης μας απασχόλησε για χρόνια. Η Σιγκαπούρη ακόμη δεν έχασε χρόνο. Περιμένουμε την ECJ και προσπαθούμε να ενημερώσουμε την συμφωνία και να μπορέσουμε και το σύστημα των επενδύσεων να το συμπεριλάβουμε εκεί. Κατανοούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαφουλεύσεις με τους ενδιαφερομένου φορείς για να δει πώς θα εφαρμογεί αυτή η συμφωνία. Εμείς είμαστε ρεαλιστές. Το πρώτο συμφέρον είναι να γίνει η επικύρωση το συντομότερο δυνατό ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν το συντομότερο δυνατό από τα ωφέλη αυτά όλες οι επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε. Θα θέλαμε να είμαστε σε στενή επαφή και όλοι ε, όσοι δεν έχουν από εσά επισκεφθεί ακόμη τη Σιγκαπούρη, σας περιμένουμε και σας καλωσορίζουμε. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και απαντήσεις. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πλήρη ανασκόπηση θα ήθελα να δώσω τώρα τον μόνιμο εισηγητή για τη Σιγκαπούρη, τον Ντέιβιτ Μάτιν, να σχολιάσει το θέμα από τη δική μας πλευρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να προσθέσω τις ευχαριστίες μου στην Υπουργό που βρίσκεται ανάμεσά μας, αλλά και για την παρουσίασή της. Χαίρομαι ιδιαίτερα που περάσαμε στην συζήτηση του περιεχομένου της ε, Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την Σιγκαπούρη. Η σημερινή συζήτηση δεν σημαίνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία κύρωση, γιατί όπω λέτε κύριε Πρόεδρε, ότι ότι καταλαβαίνουμε ότι η Επιτροπή πρότεινε δύο συμφωνίας, μία συμφωνία ελεύθερου μπορείου και μία συμφωνία διμερών ε, επενδύσεων, ελπίζω ότι θα κινηθούν ταχαίως. Το ταχαίως βεβαίως δεν είναι ένα επίρρημα που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή τη συμφωνία. Ενδεχομένω, ο Πίτερ από την Κομισιόν θα μπορούσε να μας πει πού μας εντάσσει εμάς αυτή τη διαδικασία. Τώρα, δύο πράγματα που αφορούν την ενδυνάμωση του σημείου στον οποίο αναφερθήκατε. Στην αρχή και εσείς και η υπουργό είπατε ότι οι συμφωνίες αυτές συνήθισαν το 12-13. Την ε, όταν ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αρμόδια για επενδύσεις. Ζητήσαμε από τη Σιγκαπούρη ε, να συμπεριλάμβει ένα ε, κεφάλαιο ISDS. Συμφώνησαν οι Σιγκαπούροι, είχαμε ένα κεφάλαιο ISDS, αλλά μόλις βγήκε από το σύστημα, δεν ξέραμε γιατί το θέλαμε αυτό το κεφάλαιο, και ζητήσαμε από τους Σιγκαπούριους να μας πούν αν δέχονται ένα τέτοιο σύστημα. Ε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ευχαριστώ στους Σιγκαπούριους για την υπομονή τους και την ευελιξία τους. Και αν βάλετε σε αυτό το μείγμα και το Brexit θα καταλάβετε σε τι πλαίσιο αρχίσαμε να διαπραγματευόμαστε. Όπως ε, ε, είπε και η Υπουργός, η Σιγκαπούρη είναι η πλέον σημαντική εταίρος. Και το παράδειγμα στο οποίο θέλω πάντοτε να παραθέτω είναι ότι η Σιγκαπούρη είναι ένα, μια μικρή χώρα, αλλά μετά τη Γαλλία και τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι από τις μεγαλύτερες αγοριές σκοτσέζικου ε, ουίσκι όχι γιατί πίνουν οι ίδιοι πολλοί οι κάτοικοι, αλλά γιατί είναι κέντρο διανομής. Η Υπουργό αναφέρθηκε σε μερικά από τα πλεονεκτήματα τη συμφωνία. Επιτρέψα μου, εν συντομία, να αναφερθώ σε πέντε από αυτά. Καταρχά, η συμφωνία αυτή θα μπορέσει να εξαλείψει τον χαρακτηρισμό όλων των αγαθών Εδώ μιλάμε για 51 δισεκατομμύρια. Δεύτερον, εξαλείφει όλα τα εμπόδια από το τομέα των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών και αυτός είναι ένας θετικός κατάλογος για υπηρεσίες, είναι το ΣΥΤΑ Πλάσα. Οι Σιγκαπουριανοί συμφώνησαν να προστατεύσουν ε, τις 200 ε, γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, γιατί αυτή είναι μια μονομερής παναχώρηση προς εμάς. Επίσης γνωρίζω ότι την εποχή των διαπραγματεύσεων η που είναι ενό ανέκπληξη για το γεγονό ότι δεν το έκαναν και οι Αμερικάνοι. Τώρα, τέταρτο, σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδύσεων, το ISDS ε, αντικαταστάθηκε από ένα σύστημα επενδύσεων και το άλλο, δεν ξέρω αν αυτό είναι μια βελτίωση της ε, ε, ΣΥΤΑ. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη του εμπορίου, αυτό προωθεί την σύσταση ε, μιας ομάδας TSE η οποία θα συστατεί από ανώτατους αξιωματούχους από η κοινωνία των πολιτών θα υπάρχουν συμβουλευτικές ομάδες, ομάδες ειδικών παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζω ότι έχουν κυρωθεί μόνο πέντε από τις 8 συμβάσεις και ενδεχομένως θα έπρεπε να επιτελεστεί κάποια πρόεδρος εδώ πριν περάσουμε στην επόμενη συμφωνία. Ελπίζω ότι η συμφωνία αυτή θα γίνει σύντομα και ελπίζω να μπορέσει το συντομότερο δυνατόν να περάσει από το Κοινοβούλιο. Θα ενημερώσω γι' αυτό και τους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είμαστε πριν από το Χριστούγεννα και είναι πλέον πρόσφορη η εποχή για να ελπίζουμε. Ο κύριος Χάμπακ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας βλέπουμε στις σχετικά κρύες Βρυξέλλες. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα μπορούσα να μιλήσω εξ ονόματος της ομάδας του ΕΛΚ δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ήδη ο εισηγητής, το πόσο καλά προετοιμασμένη είναι αυτή η εμπορική συμφωνία. Βεβαίως η Σιγκαπούρη ήταν ένας πάρα πολύ καλός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουμε ότι αυτή η εμπορική συμφωνία θα πρέπει να συναυθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για κάτι, κάποια καθυστέρηση από πλευρά τη ευρωπαϊκή Ένωσης γιατί δεν είναι εύκολο να βρεθούν γύρω από το ίδιο το τραπέζι τόσες πολλές ε, χώρες. Εδώ βρισκόμαστε 28 χώρες, αλλά χρειάζεται χρόνος για όλα αυτά. Το ΕΛΚ βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, πίσω από αυτή την εμπορική συμφωνία και πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε πολύ περισσότερα του χρόνου και στις δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και περιμένουμε με ανυπομονησία αυτή τη συμφωνία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλώς κύριε Υπουργέ. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κατανόηση που δείχνετε με τα εσωτερικά συστήματα που έχουμε. Μεγάλη μου χαρά που σας βλέπω εδώ σήμερα και ελπίζω όλοι εδώ σε αυτή την ε, αίθουσα θα στείλουν το μήνυμα ότι θα πρέπει να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία έτσι ώστε και οι καταναλωτές να μπορούσαν να, να την εκμεταλλευτούν και πραγματικά έχουμε σοβαρές αντιρρήσεις σε οποιαδήποτε προσπάθεια να ανοίξει και πάλι αυτή η συμφωνία. θα πρέπει να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις των εμπορικών μας εταίρων στη Σιγκαπούρη. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα τώρα προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά της ε, Σιγκαπούρης. Θα ήθελα να γνωρίζω αν υπήρξε μια περαιτέρω καθυστέρηση και αν υπήρξε, αυτό θα επηρέαζε πρακτικά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω την Επιτροπή που μας ακούει. Τι κάνει η Επιτροπή για να τα προωθήσει όλα αυτά, για να αυξηθεί η γνώση και η ευαισθησία για αυτή την ε, συμφωνία, για να μπορέσει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε την Υπουργό για την παρουσία της εδώ. Οι διαπραγματεύσεις ε, με τη Σιγκαπούρη ολοκληρώθηκαν ήδη από το 2014 και έκτοτε ε, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολήθηκε με την έκδοση μιας γνωμοδότησης σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί αυτής της συμφωνίας και βέβαια αυτή η κατάσταση μας ε, δυσκολεύει. Γιατί δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή μια αξιολόγηση αντικτύπου σε ό,τι αφορά τη σύναψη μια τέτοια συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Ε, η σχετική αξιολόγηση αντικτύπου για την ΑΖΕΑΝ συντάχθηκε το 2009. Αλλά βέβαια υπάρχει ετερογένεια μεταξύ των χωρών τη ΑΖΕΑΝ. Διαφορετική η Σιγκαπούρη από τη Μαλαισία και διαφορετική η Μαλαισία από τι Φιλιππίνε. Και βέβαια οι διαφορέ μεταξύ των χωρών τη ΑΖΕΑΝ είναι μεγαλύτερε από ό,τι για παράδειγμα μεταξύ τη Γερμανία ε, ε, και τη Ελλάδα ή μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οπότε από εκεί και μετά έχουν συμβεί και διάφορα από το 2009, δηλαδή από την εκπόνηση τη τελευταία τελευταία αξιολογή που Τότε προσπαθούσαμε να βγούμε από την τραπεζική κρίση. Έκτοτε έχουμε καταφέρει να λύσουμε τα διδάγματά μα σε ό,τι αφορά και την ε, ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, την ε, συγκέντρωση των ε, για τι συγχωνεύσεις των ε, τραπεζών και ούτω καθεξής. Οπότε θα ήθελα να υπάρξει μια αξιολόγηση και μια ανάλυση ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο για την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Δεν ξέρω δηλαδή ποιε θα είναι τελικά οι επιπτώσεις ε, ε, μια τέτοια συμφωνίας για την οικονομική σταθερότητα τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και της Σιγκαπούρη. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ σημαντικό εμπορικό εταιρό όταν αναφερόμαστε στη Σιγκαπούρη και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη Σιγκαπούρη ω προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μια τόσο βαθιά και περιεκτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης θα μπορούσε πράγματι να έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, στις ε, ε, οικονομίες μας αλλά και στις κοινωνίες μας και στο κανονιστικό μας πλαίσιο και κατά συνέπεια θα έπρεπε να προβλέψουμε κάτι σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό, το κανονιστικό πλαίσιο ποια δηλαδή θα είναι τα, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας προκειμένου να διασφαλίζουν την οικονομική σταθερότητα Δηλαδή η οικονομική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Σιγκαπούρη θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενό διαφορετικού θεσμικού πλαισίου. Τι θα συμβαίνει για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των ε, ε, επενδύσεων. Εδώ ανέφερε το δικαστήριο ότι αυτό το ζήτημα θα περιλαμβάνει τη συναρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό τι σημαίνει ότι το σχετικό κεφάλαιο θα εξαιρεθεί εντελώ από τη συμφωνία. Η ε, ε, Επίτροπο Μάστρομ ανέφερε πρόσφατα ότι η Όποιε διαφοροποιήσει ε, που θα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτές τις συμφωνίες ε, μελλοντικά δεν θα αποτελούν πλέον αντικείμενο εξέταση από την πλευρά του δικαστηρίου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι οι επενδύσει και οι συμφωνίε επί επενδύσεων θα είναι εντελώ ξεχωριστέ και δεν θα περιλαμβάνονται πλέον σε τέτοιου είδου συμφωνίε. και σε σχέση με αυτό θα ήθελα να ακούσω και ένα σχόλιο από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Πίτερ από την πλευρά της Επιτροπής ε, βρίσκεται σήμερα εδώ, οπότε ελπίζω πως ε, θα δώσετε κάποιες απαντήσεις. Η ε, Γιούτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Ήδη έχουν υποθεί πολλά. Εγώ θα, κατά βάση πιστεύω ότι λίγο σας κοροϊδέψαμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πραγματικά μας βάζει σε μια δύσκολη θέση τώρα που βρισκόμαστε σε φάση λεπτομερούς εξέτασης του περιεχομένου της ε, συμφωνίας. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει μια δημοκρατική συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά με το πώς θα αναπτυχθεί αυτή η πολιτική. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την υπομονή σας. Θα μπορούσαμε τώρα να ασχοληθούμε με το περιεχόμενο της συμφωνίας υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δεν αναλύθηκαν επαρκώς. Αυτό που θέλουμε που μας ε, απασχολεί είναι το θέμα της κύρωσης των συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η, Συγκαφέ, Σιγκαπούρη δεν έχει κυρώσει τρεις ε, από αυτές. Η τρίτη αφορά την ε, ε, ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Εκεί είναι λίγο προβληματικός ο τρόπος ε, ε, της οργάνωσης των συνδικάτων και της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε αν θα ήσασταν διατεθειμένοι στο χρόνο που απομένει να ξεκινήσετε ένα διάλογο σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα εφαρμοστούν οι αρχές που βρίσκονται εδώ. Αυτό δεν αφορά μόνο τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης. Θα πρέπει η συμφωνία να τεθεί σε ένα γενικότερο ε, πλαίσιο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές τάσεις προστατευτισμού. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η γενική διακυβέρνηση, η παγκόσμια διακυβέρνηση και να δούμε ποια είναι η υποστήριξη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Με απασχόλησε λίγο θα έλεγα όταν είδα ότι φέτος η Επιτροπή οποίοι Εμπειρογνωμόνων ε, ζήτησαν την άποψη της Σιγκαπούρης για θέματα εφαρμογής ε, ε, στον τομέα της εργασίας, των προτύπων εργασίας. Το θέμα είναι το πώς θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε για να αναπτύξουμε ένα διάλογο και να έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλες αυτές οι δεσμεύσεις θα μεταγραφούν και πρακτικά και αυτό σε ό,τι αφορά και τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Υπουργό που είναι παρούσα και να αναγνωρίσω την εργασία που επιτελέσατε και εσείς εκπροσωπώντας την κυβέρνησή σας. Όπως είπαν οι συνάδελφοι και Ζουτ, όλες οι καθυστερήσεις που έγιναν έγιναν δεδομένου ότι ήθελε να κάνει την εργασία του σωστά και η κυβέρνηση και εμείς, αλλά οι καθυστερήσεις επειδή υπήρχαν νομικά προβλήματα και άλλα δικαιολογούνταν γιατί είναι σημαντικά τα θέματα. Θα ήθελα να πω το εξής. Υπογραμμίστηκαν όλες οι θετικές πλευρές αυτής της συμφωνίας, τις ημερίζομαι αυτά τα οποία λέχθησαν. Εγώ μπόρεσα να πάω και στην Σιγκαπούρο, και να δω επιτόπου την μεγάλη πρόοδο που υπάρχει στην χώρα αυτή. Και θα ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά ε, την, ε, ε, την, το δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης μεταξύ 188 χωρών είναι πέμπτη χώρα η Σιγκαπούρο. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε η Σιγκαπούρη δεν έχει επικυρώσει κάποιες συμφωνίες στα πλαίσια του Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας όταν χρειάστηκε να το κάνουμε. Ε, τι έχει γίνει στο μεταξύ διάστημα. Κυρίως ο όταν ε, έχουμε να κάνουμε με τη συγκεκριμένη συμφωνία και με άλλους. Για ποιο λόγο λοιπόν η Σιγκαπούρη που έχει τέτοιου είδους δείκτη που, ε, ε, τεχνολογικής οικονομικής ανάπτυξης και δείκτη ε, ανάπτυξης των πολιτών του, γιατί δεν έχει υπογράψει και επικυρώσει αυτές τις συμφωνίες, για ποιους λόγους. Και Βεβαίω για να μπορέσει να επιληθεί το όλο θέμα, τι είδου συμβαστική λύση προτείνετε εσεί. Σα ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Έχετε τώρα την δυνατότητα να απαντήσετε. the speakers ευχαριστώ. πολύ. Ευχαριστώ πολύ τα σχόλιά σας για την παρουσίασή μου. Μερικά από τα σχόλια που έγιναν, θα ήταν καλύτερο να γίνουν στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Για την ώρα όμως θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα που αναφέρθηκε σε αρκετές από τις παρεμβάσεις και που αφορά την βιωσιμότητα του εμπορίου και της εργασίας. Επιτρέψτε μου επίσης να μοιραστώ με τα παραόντα μέλη τον τρόπο με τον οποίο η Σιγκαπούρη προσεγγίζει το θέμα της προστασίας εργασίας. Υιοθετήσαμε μία τριμερή προσέγγιση η οποία αναφέρεται σε μία πολύ στενή σχέση εργασίας μεταξύ των εργαζομένων που εκπροσωπούν από τα συνδικάτα, των εργοδοτών και της κυβέρνησης. Και υπάρχει μία σειρά ε, Ε, θα πρέπει λίγο να προωθήσουμε την εργασιμότητα όλων των εργαζομένων, τη δυνατή, την απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων. Να δούμε τους νόμους που επηρεάζουν την οικονομία και τις θέσεις εργασίας. Αυτά είναι θέματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Θα μπορούσα να πω ότι αναμένεται πολλά μέλη του Κοινοβουλίου του γομετός όπου είναι στη κυβέρνηση τώρα να συνεργάζονται στενά με τα συνδικάτα. Και αυτό αφορά μια πολύ στενή σχέση. Αυτή η στενή συνεργασία μεταξύ των συνδικάτων, των εργοδοτών και της κυβέρνησης βοηθάει στην διαμόρφωση πολύ καλών θετικών αποτελεσμάτων. Κρατήσαμε την ε, ανεργία σε χαμηλό επίπεδο στο 3% και το ποσοστό απασχολησιμότητας ε, ακολούθησε μία ανωδική τάση και ξεπέρασε το 65% το 2016. Υπάρχει και αυτή η προσέγγιση που μας επιτρέπει διαρκώς να ζητάμε αυξήσεις ημερομισθείων για τους εργαζόμενους. Και πιστεύω, όπως είπε και ένας από τους ομιλητές, αυτή είναι μια συγκεκριμένη προσέγγιση και αυτό θα πρέπει να πω ότι συνέβαλε στο να βελτιώσει τη γενικότερη απόδοσή μας ό,τι αφορά άλλα θέματα. Η Σιγκαπούρη τα πήγε καλά. Ε, είτε μιλάμε για υπηρεσίες, είτε για οτιδήποτε άλλο. Επίσης έχουμε στενή σχέση με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους και συνδιοργανώνουμε ε, διάφορες ε, διοργανώσεις προκειμένου να συζητηθούν μερικές ε, εργασιακές πρακτικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσέγγισή μας για τις συμβάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι παίρνουμε, λαμβάνουμε σοβαρά την προσχώρησή μας στις συμβάσεις και πριν το κάνουμε αυτό θέλουμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να συμμορφωθούμε και με το γράμμα και με το πνεύμα της σύμβασης. Παρόλα αυτά επανεξετάζουμε τους εγχώριους νόμους και κανονισμούς με στόχο να τους ευθυγραμμίσουμε περισσότερο με το περιεχόμενο των συμβάσεων. Και δίχως άλλο, με πολύ μεγάλη χαρά, συνεχίζουμε να είμαστε σε επαφή με τα μέλη και όπως είπε πρόσφατα η κυρία Κατεντάλε, ξεκινάμε ένα διάλογο για να μπορέσουμε να δείξουμε στα μέλη πώς ε, η τριμερής αυτή αντίληψη βοηθάει στην αύξηση των ημερομυστίων και της απασχολησιμότητας στη Σιγκαπούρη. Και για ποιο λόγο ακριβώς εμείς υποστηρίζουμε τον περιεχόμενο όλων των συμβάσεων, των βασικών συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Thanks a lot, ε, Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Τώρα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσουμε τον λόγο στον πολύ γνωστό Πίτερ Μπέατς, ο οποίος είναι αρμόδιος ε, για μία σειρά από χώρες εκεί, Νοτιοανατολική Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, και ούτω καθεξής, Πρόεδρε, και άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ, ε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ μέλη εδώ της Επιτροπής. Ε, πράγματι πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία με ένα σημαντικό συμπορικό εταίρο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβω τη σημασία αυτής της ε, οικονομικής μας ε, σχέσης. Νομίζω πως την εξέθεσε αναλυτικά η υπουργό και νομίζω πως η συμφωνία με την Σιγκαπούριο ήταν η πρώτη η οποία συνήφθη με ένα μέλος της ΑΖΕΑΝ Προσπαθήσαμε βέβαια να συνάψουμε με τέτοια συμφωνία από το 2007 έως το 2009 με την ίδια την ΑΖΕΑΝ και ε, από εκεί και μετά ξεκινήσαμε δίμερες διαπραγματεύσεις με πρώτη αυτήν εδώ και ελπίζουμε ότι θα δώσει συνέχεια σε μια σειρά από άλλες διμερείς συμφωνίες. Ε. Από εκεί και μετά πρόκειται για μια ε, συνολική προσέγγιση που έχουμε με τις χώρες της ε, περιοχής. Έχουμε μια πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κορέα και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και πολλές ακόμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εδραιώνουμε την παρουσία μας στην περιοχή και αξιώνουμε και την αξιοπιστία της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης στην Ασία. Πρόκειται επίσης και για την πιο φιλόδοξη και περιεκτική συμφωνία την οποία έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια χώρα της Ασίας και ειδικότερα δε με μια χώρα της ΑΖΕΑ. Ε, γι' αυτόν τον λόγο και η Επίτροπος αποφάσισε να δώσει μια σημαντική ομιλία σε σχέση με τη Σιγκαπούρη νωρίτερα φέτο, ε, όπου επιβεβαίωσε ακριβώ τη βούλησή μα να ενισχύσουμε τι εμπορικέ μα ε, σχέσει με του εμπορικού μα εταίρου στην Ασία. Μετά από την προσαρμογή των ε, διατάξεων σε ό,τι αφορά τι επενδύσει το 7 η συμφωνία περιλαμβάνει και το μηχανισμό επίλυση διαφορών και τι επενδύσει με όλε τι ε, βελτιώσει, οι οποίε ακόμα ε, δεν έχουν ε, για παράδειγμα ληφθεί ακόμα υπόψη στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών. Αναμένουμε λοιπόν την ταχύτερη δυνατή εφαρμογή στην πράξη αυτής της αναδιαπραγματευμένης συμφωνία. και συμμεριζόμαστε λοιπόν αυτήν την ελπίδα τη δική σα επιτροπή για την ταχεία θέση σε ισχύ και επιχαίρουμε το γεγονός ότι ήδη έχει προβαίνει σε ανταλλαγή απόψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα ζητήματα χωρίς να έχει ακόμα υποβληθεί επισήμω το Κοινοβούλιο συγκεκριμένη συμφωνία για να δώσει την έγκρισή του. Μετά από την έκδοση και τη απόφαση από την πλευρά του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αρμοδιότητα, είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί ενεργά επί των ζητημάτων των ε, Συμφωνιών Ελευθερίου Εμπορίου και ε, πράγματι τα ψηφίσματα σε ό,τι αφορά ε, τι διαπραγματευτικέ εντολέ για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, αλλά και οι συγκεκριμένε τοποθετήσει του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τη μελλοντική αρχιτεκτονική τέτοιου είδου συμφωνιών είναι σημαντικά. Ε, καθώς οριστικοποιούμε λοιπόν το συγκεκριμένο κείμενο και τις ε, μεταφράσεις του στις διάφορες γλώσσες που βέβαια χρειάζονται χρόνο, συνεχίζουμε να είμαστε σε επαφή με τα κρατη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική, τη δομή τόσο αυτής όσο και των υπολείπων μελλοντικών συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και επενδύσεων. Αλλά σίγουρα έχουν γίνει ήδη πολλά έτσι ώστε να προετοιμάσουμε, να προπαρασκευάσουμε την εφαρμογή της συμφωνίας στην πράξη. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα τεθεί σε ισχύ ε, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως και από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητε outreach και γενικότερη επαφή και ευαισθητοποίηση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία έτσι ώστε όλοι οι αρμόδιοι φορεί, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί να γνωρίζουν ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουμε από αυτή τη συμφωνία έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό για λόγο συμφωνία. Αναμένω με ενδιαφέρον τι περισσότερε ανταλλαγέ απόψεων που θα ακολουθήσουν με την Επιτροπή σα και στο πλαίσιο τη εντολή που θα δοθεί αργότερα σε ό,τι αφορά δηλαδή, και την έγκριση από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Και αυτά από την ε, πλευρά μου, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, και ε, ο κύριο Ντέβιτ Μάρτινο, ο μα, θα πάρει το λόγο για τα καταλακτικά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, Έμα, να πω ότι νομίζω κανεί δεν είναι υπέρ του να ξανανοίξουν οι διαπραγματεύσει επί τη συμφωνία. Νομίζω πω έχουν ολοκληρωθεί αυτέ οι διαπραγματεύσει και ε, η Σιγκαπούρη υπήρξε πολύ υπομονετική σε ό,τι αφορά τι δικέ μα καθυστερήσει. Οπότε δεν νομίζω πω υπάρχει κανένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να θέλει να αναδιαπραγματευτούμε αυτή τη συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά όπω είπαν και οι ε, ακόμα και σε σχέση με τον Καναδά, όπου έχουμε μια, ένα όριμο δημοκρατικό ε, συνεχίσαμε να επιμένουμε σε ό,τι αφορά την εκύρωση των συμφωνιών του ΆΕΛΟ που δεν είχαν υπογραφεί ακόμα. Οπότε ελπίζω πω ε, θα υπάρξει και αντίστοιχη πρόοδο από την δική σα πλευρά. Βέβαια, είναι στενό το χρονοδιάγραμμα, οπότε δεν ε, περιμένω ότι πράγματι θα έχουν ε, κυρωθεί μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας μας εν λόγω ε, ε, συμφωνίες του ΑΕΛΟ, αλλά αναμένουμε μια δέσμευση από την πλευρά της Σιγκαπούρης ότι θα το πράξει στο μέλλον. Και επιτρέψτε μου επίση να πω, για να σημειωθεί στα πρακτικά, ότι εσεί ως Σιγκαπούρη, σε αντίθεση με άλλε γειτονικέ σα χώρε, πραγματικά είστε ένα κράτο δικαίου. Δηλαδή, όταν, όταν κυρώνεται μια συμφωνία την εφαρμόζετε στην πράξη σε αντίθεση με άλλε γειτονικέ σα ε, χώρε οι οποίε δεν το κάνουν. Οπότε ε, πραγματικά αντιλαμβανόμαστε του περιορισμού σα, αλλά η ε, κύρωση τη συμφωνία από την πλευρά του Κοινοβουλίου θα ήταν πολύ ευκολότερη αν είχαμε το μήνυμα από εσά ότι θα προβείτε στην κύρωση των τριών υπολοιπόμενων συμφωνιών ε, τη Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα όσα ανέφερε ο Πίτερ από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πω ότι αναμένω ότι ελπίζω τα κράτη-μέλη που είχαν κάποιες επιφυλάξεις σε συνέχεια της απόφασης ε, που εξέδωσε το δικαστήριο να ε, κυρώσουν από την πλευρά τους και μάλιστα το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Καλώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, σε σχέση ουσιαστικά με αυτές τις δύο συμφωνίες. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά κυρία Υπουργέ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να ατηρώσουμε στις αρχές του επόμενου έτους αυτή τη συμφωνία. So, dear Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο μας θέμα, το 9 ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινή εμπορικής πολιτικής. Η συγγήτρια, η κυρία Σαϊφή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή τη στιγμή εκπονώ την ε, σχέδιο έκθεσης για την ε, κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα σήμερα να κάνω μια πρώτη παρατήρηση για να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Τα πλαίσια με στο οποίο κινούμεθα άλλαξε από τότε που εμφανίστηκε το 2015 το έγγραφο της κοινή στρατηγικής. Οι ΙΠΑ βρίσκονται σε κάποιος ε, ε, οπισθοδρομική θέση. Το Brexit αυτή τη στιγμή το διαπραγματευόμαστε. Η ψηφιοποίηση προχωρεί με μεγάλη ταχύτητα και δίθενται πάρα πολλά ερωτήματα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής. Γι' αυτό η στρατηγική της κοινή εμπορικής πολιτικής ε, ε, στην, ε, στη μέση χρονική περίοδο είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις από κοινού. Πρώτα απ' όλα, ως πρώτη εμπορική δύναμη να το κόσμο θα πρέπει να μπορούμε ακόμη περισσότερο να προσβλέπουμε στην προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών και των επιχειρητήσεων για να μπορέσουμε να προασπίσουμε τις αρχές της δικαίου εμπορίου βάσει αρχών που θα γίνονται σεβαστές από όλους και με και με αρχές κλειδιά όπως αυτή της αμοιβαιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ισοσκελισμένες συμφωνίες και να θεσπίσουμε μέτρα για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε τον ε, αθέμητο ανταγωνισμό στα πλαίσια των συντονισμένων προσπαθειών που κάνουμε στα πλαίσια όλων των κοινών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτής της κοινή εμπορικής πολιτικής πρέπει να πω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είναι λοιπόν σημαντικό το περιεχόμενο των συμφωνιών να εφαρμοστεί και τα ευρωπαϊκά εργαλεία και μέσα που διαθέτουμε να χρησιμοποιηθούν πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ανακοίνωση μεταξύ όλων των μέσων τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με ποιος θα χρησιμοποιηθεί. Η εργασία με τις πρεσβείες και με όλους τους υπεύθυνου φορείς είναι προ... Αρχική σημασία και θα πρέπει να υπάρχει όχι μόνο όταν γίνεται διαπραγμάτευση συμφωνιών, αλλά και μετά κατά την περίοδο παρακολούθηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτό από την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή αυτών των ε, εμποριών θα μπορούσε μέσα στα έναν ευρωπαϊκό ε, οδικό χάρτη να μας πει που βρίσκεται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε συμφωνία. Η εμπορική μας κοινή πολιτική θα πρέπει να ενισχύει και να προγάγει κυρίως τα συμφέροντα και τις αρχές μας. Να λαμβάνουμε υπόψη τις γενικευμένες προτιμήσεις σε όλα τα πλαίσια ε, των πολιτικών μας να είμαστε προσεκτικοί ώστε στον ε, τομέα τον κοινωνικό και της προσοχής του περιβάλλοντος να είμαστε οι καλύτεροι παγκοσμίω και κυρίως να προσθέτουμε τους εργαζόμενους. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι η διαφάνεια είναι πρωταρχική σημασία. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν ποια είναι τα συν και τα πλην κάθε συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε διαφάνεια από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει λοιπόν να έχει καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική, κυρίως όσον αφορά τις μελέτες αντικτύπου και τα αποτελέσματα. Και να είναι ο ε, φορέας που θα συνδέσει τι διάφορε συζητήσει που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα Εθνικά Κοινοβούλια και στα κράτη-μέλη. Είναι ευρύτατο το θέμα αυτό και χαίρομαι που σήμερα αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα μα βοηθήσει να προχωρήσουμε και μεγάλη ευχαρίστηση θα ακούσω όλα τα σχόλια που θα υποβάλλετε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Σαϊφή. Δίνω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Κύριε Ντάλητα πρώτη, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαϊφή Συμφωνώ απολύτως με πολλά από τα σημεία τα οποία υπογράμμισε αρχίζοντας πέρσι, νομίζω. Είδαμε το άλλο θέμα να και ξέρουμε ότι η εμπορική μας πολιτική και η εμπορική η κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πέρσι έχουν διαγράψει μεγάλες αλλαγές. Και εξελίσσαν τα πράγματα και νομίζω ότι έχουμε πρόσφατα δημοσίευση της έκθεσης για τις FTAs που μας δίνει συγκεκριμένα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε για να δούμε πώς θα εφαρμογεί στην πράξη η κοινή εμπορική πολιτική. Παρά το γεγονός ότι χαιρετήσαμε αυτή την έκθεση και είναι η πρώτη ε, φορά που δημοσιεύεται αυτή η έκθεση επί της εφαρμογής πρέπει να πω ότι δεν έχει ένα περιεχόμενο το οποίο ίσως δεν είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Είναι πολύ ε, αισιόδοξο διότι παρουσιάζονται ρόδινα μέσα από τις στατιστικές και δεν υπάρχει εξοσκελισμένη προσέγγιση μεταξύ του θετικού και αρνητικού αντικτύπου της εφαρμογής αυτής της ε, κοινή εμπορική πολιτική. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να παρουσιάζουμε αντικειμενικά όλα τα στοιχεία όταν μιλούμε για εφαρμογή. Και είναι δύσκολο να είναι κανείς ίσως πάντα πολύ αντικειμενικός. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν ε, κάποιες μονομερείς απόψεις. Μας παρουσιάζει κάποιες επιτυχείς ιστορίες τομέων επιχειρήσεων. Στον εμπορικό τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να μιλάει ότι σε κάποιους τομείς, να λέγει ότι σε κάποιους τομείς χάνονται θέσεις απασχόλησης, μεταφέρονται επιχειρήσεις, μεταφέρονται θέσεις απασχόλησης, για να δώσω ένα παράδειγμα, και δεν αναφέρει και πολύ τον αντίπτυπο της κοινή εμπορικής πολιτικής γενικότερα στην ε, σφαιρική οικονομική ανάπτυξη. Όταν βλέπουμε λοιπόν πώς ε, τα FTS εφαρμόζονται, δεν βλέπουμε τον αντίκτυπο για τις χώρες ευρωπαϊκές. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό να το έχουμε κατά νου και να το γνωρίζουμε ως στοιχείο. Όπως είπε και η κυρία Σαφή, υπάρχουν θέματα αξιών και θέματα που αφορούν το πώς αναπτύσσεται και πώς εφαρμόζεται στην πράξη η πολιτική μας αυτή. Εξετάζοντας λοιπόν αυτή την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσα ότι πολύ λίγοι από τους κανόνες που υιοθετούνται στον τομέα αυτό εφαρμόζονται στην πράξη. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το μελετήσουμε περαιτέρω. Για τις ε, ε, θέματα στα θέμα σταδιοδρομιών που υπάρχει στον τομέα αυτό, εξετάζοντας τι ακριβώς ε, γίνεται με την έκθεση της Επιτροπής. Λίγα λέγονται για τις κρατικές ε, επιχειρήσεις, για την ε, συμμετοχή κάποιων μεν Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κοινά. Θα πρέπει να την συζητήσουμε τη έκθεση αυτή για να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια ισορροπημένη άποψη για την κοινή εμπορική πολιτική. Και συμφωνώ με την τελευταία παρατήρηση κυρία Σαφή. Είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια Μόνον έτσι και μόνο όταν έχουμε μία αντικειμενική και σαφή άποψη για την εμπορική μας πολιτική με πλήρη διαφάνεια θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών και να είμαστε σίγουροι ότι ε, προωθούμε μία πολιτική προς όφελος όλων και όχι προς το συμφέρον ολίγων. Ευχαριστώ. Μιλάω εξ ονόματος του σχεδίου εισηγητή Ζάντο, εμείς προσπαθούμε να προκύψουν συγκεκριμένα ωφέλη για την οικονομία και τους ανθρώπους. Πρόσφατα ε, ολοκληρώθηκε η Συμφωνία με τη το Καναδά, την, την Ιαπωνία, ε, το Περού και η φάση της εφαρμογής είναι σημαντική. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των ε, συμφωνιών στις επιχειρήσεις. θα θέλαμε να δούμε ότι είναι μία ε, πρακτική προσέγγιση. Δεν θα είναι εύκολη άσκηση γιατί η ε, όλα αυτά έχουν σχέση με τις φιλοδοξίες μας. Ε, και βεβαίως διαφέρουν και οι φιλοδοξίες μας παρόλα αυτά. Συμφωνήσαμε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και συγκεκριμένοι προσανατολισμοί. Και αυτή είναι μια παράλληλη διαδικασία. Αυτές οι δύο διαδικασίες θα πρέπει να γεννηθούν παράλληλα. Στην αρχική φάση θα ήθελα να αναφερθώ στα ερωτήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ένα, οι εταιρείε Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν εκμεταλλεύονται την ευκαιρία που τους παρέχεται. Για ποιο λόγο οι εταιρείε Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το 70% των επιλέξιμων εξαγωγών. Οι εταίροι μας χρησιμοποιούν το 90%. Πώς θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε ε, μια μεγαλύτερη εκμετάλλευση των ευκαιριών. Θα πρέπει να μας απασχολήσει το πώς ε, ε, θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Τι είδους στρατηγικές επικοινωνίας είναι αναγκαίες. Δύο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που αφορούν το 30% των εξαγωγών βρίσκονται αντιμέτωπες με πάρα πολλές προκλήσεις. Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά αποτελούν θέματα των διαπραγματεύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα αναζητήσει αυτά κεφάλαια Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να κοιτάξουμε τη διαδικασία αυτή προκειμένου να υπάρξει η αύξηση της συμμετοχής περαιτέρω. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν ε, άρδιν τα μοντέλα τους. υπάρχει θα πρέπει να υπάρξει πρόσβαση στις ε, διεθνείς ε, αγορές. Θα, πρέπει όμως πρέπει να βασιστούμε στη τεχνολογία και χρησιμοποιώντας τους ε, διάβλους διανομής. Θα πρέπει να υπάρξει διαφορερά στις στρατηγικές. Θα πρέπει να δοθεί βοήθεια στο εμπόριο θα πρέπει να αυξήσουμε την δυνατότητα των αναπτυσσόμενων χωρών για να προωθηθεί η συμφωνία ε, στη ε, ε, εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε υπέρ του να οδηγηθούμε σε μια απτή ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες. Θα πρέπει να βρούμε καινοτόμους τρόπους και να αναπτύξουμε περισσότερες συνέργειες και η πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι ζητάμε σεβασμό στους εταίρους μας σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βεβαίως υπάρχουν και οι δεσμεύσεις μας. Είναι απόλυτα σημαντικό να ενδυναμώσουμε όλα αυτά. Θα ήθελα όμως, ε, δεν θα ήθελα η σημαντική αυτή έκθεση να παρασυρθεί από το θέμα της όπως έγινε στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Βέβαια πολύ απέχουμε από τα συμπεράσματα παρόλα αυτά εγώ ήθελα να προειδοποιήσω. Με ανυπομονησία περιμένω να δω την έκθεση. Ευχαριστούμε ε, για τους, ε, τους ε, φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συμφωνήσω με την εισηγήτρια σε σχέση με τα όσα είπε ε, κατά την σχόλιά της ότι δηλαδή το περιβάλλον έχει μεταβληθεί εντελώς και κατά συνέπεια θα πρέπει να τα αποκριθούμε σε αυτό το νέο περιβάλλον. Εάν λάβουμε υπόψη μας δηλαδή την τοποθέτηση ε, της Αμερικής για παράδειγμα όχι μόνο απέναντί μας αλλά και στο πλαίσιο της TIP, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, νομίζω πως δημιουργείται η δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εφαρμόσει μια φιλελεύθερη εμπορική πολιτική. Οπότε θα ήθελα η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει εδώ την πρωτοβουλία, να αναζητήσει νέες αγορές, αλλά ταυτόχρονα, όπως ήδη αναφέρθηκε, να δει το τι μπορεί να κάνει σε σχέση με τους υφιστάμενους εμπορικούς μας εταίρους. Για παράδειγμα, εξυγχρονίζοντας τις υφιστάμενες συμφωνίες, αλλά και στο επίπεδο της εφαρμογής των υφιστάμενων ε, ε, εμπορικών συμφωνιών. Άρα λοιπόν νομίζω πως σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οθετήσει την ε, ε, σωστή προσέγγιση, δηλαδή αναζητώντας νέους εμπορικούς εταίρους και ολοκληρώνοντας τις συμφωνίες με εταίρους οι οποίοι επιθυμούν να υπάρχει ένα πολυμερές, ένα προοδευτικό σύστημα που θα βασίζεται σε συγκεκριμένου κανόνες. Και αυτό με φέρνει σε μια ακόμα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να συνεχίσει να επιέζει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας για την εφαρμογή ενός πολυμερού συστήματος εμπορικών ορίο που θα βασίζεται σε κανόνε. Επίση, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τι συμφωνίε μα έτσι ώστε να περιλαμβάνουν ε, νέου κλάδου οι οποίοι σχετίζονται περισσότερο με το εμπόριο σήμερα. Γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει ω προ το ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί κλάδοι κλειδιά. Για παράδειγμα, θα πρέπει να περιλάβουμε σε όλε τι μελλοντικέ μα συμφωνίε και ένα κεφάλαιο σε ό,τι αφορά το ψηφιακό εμπόριο, έτσι ώστε να καλύψουμε εκεί μεταξύ άλλων και τι ροέ των δεδομένων. Κλείνοντα, να αναφερθώ σε κάτι που αναφέρατε κι εσείς ε, κύριε Συγήτρια και με το οποίο συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν αποτελέσματα αυτά για τις επιχειρήσεις μας, για τις οικονομίες μας, για τους πολίτες μας αλλά θα πρέπει να καταστήσουμε και ορατά, δηλαδή γνωστά αυτά τα θετικά αποτελέσματα σε αυτούς τους ε, πολίτες αυτές τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος ε, και την ο Helmut Scholz έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ευκαιρία που μας δίδεται ίσως μια φορά το χρόνο να εξετάζουμε πιο λεπτομεριακά το θέμα της εφαρμογής κοινή εμπορικής πολιτικής. Λέγουν όλοι οι συνάδελφοι ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τα τεκνενόμενα, τις ε, ε, αλλαγές, τα μέσα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να θέτουμε σε εφαρμογή την κοινή εμπορική πολιτική. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε και τα προβλήματα, τα μειονεκτήματα, τα κενά και όχι μόνο τα θετικά. Και βεβαίως εδώ πρέπει να αντιμετωπίζουμε και την πολυπλοκότητα της σύγχρονης οικονομικής ζωής, της οποίας η εμπορική πολιτική είναι μόνο μία πτυχή. Στην ε, έκθεση το 2015 για πρώτη φορά παρουσιάστηκε η ιδέα αυτή των ε, ε δυνατότητας εκπόνηση ετησίων εκθέσεων, πράγμα που είναι θετικό. Θα ήθελα να κάνω τρεις συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Και βεβαίως προσβλέπω σε συνεργασία με την εισηγήτρια. Πρόσφατα στην Επιτροπή μας συζητήσαμε την οικονομική διακυβέρνηση του τομέα του εμπορίου. Και το ερώτημα είναι όταν μιλούμε για κανόνες που πρέπει να ισχύουν και στους οποίους να βασίζεται η εμπορική μας πολιτική θα πρέπει να συμπεριλάγουμε και για το ποιος θέτει αυτούς τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουμε. Ποιος τους ορίζει. Διότι εφαρμογή ε, της πολιτικής αυτής και οι εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να αναφέρουν και ποιοι υποφελούνται από αυτή την εμπορική πολιτική την κίνη. Διότι εμείς αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε μόνο για να προωθήσουμε το εμπόριο, για να προωθήσουμε όμως γενικότερα τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς όφελος των πολιτών μας. Το επόμενο θέμα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ε, ε, εποπτεία των ε, άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων και μέσων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του εμπορίου και γενικότερα για την οικονομική ανάπτυξη. Και με μεγάλη προσοχή να εξετάζουμε την ε, οριζόντια σχέση μεταξύ των διαφόρων εμπορικών συμφωνιών και να δούμε ποιο είναι το σορευτικό αποτέλεσμα μία συμφωνίας στην άλλη. Πάντα λοιπόν μαθαίνουμε από αυτό το οποίο γίνεται. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν Τι ακριβώς συμβαίνει στα πλαίσια των νέων στρατηγικών που πρέπει να αναπτύξουν. Σας ευχαριστούμε και για τους απράσινους ο κύριος Μπούχνα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια για τα πολύ καλά ρεθίσματα για σκέψη που μας έδωσε. Ε, αλλά θα ήθελα να παίξω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου σήμερα κατά τη δική μου άποψη αυτή η έκθεση της ε, Επιτροπής είναι θετικό το ότι περιλαμβάνει ήδη κάποια ε, κριτικά σχόλια, επικριτικά σχόλια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Μεξικό και τη συγκεκριμένη συμφωνία και το τι αυτή θα σημάνει σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχεια, ε, θα μπορούσε να έχει σημάνει την καταπολέμηση της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, πολλά θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αν είχαμε προβεί σε διαφορετικού είδους διαπραγματεύσεις. Ήδη δηλαδή ε, ξέραμε ε, ήδη κάποια εντύπωση ως προς το πώς θα πήγαιναν τα πράγματα αφού είχαμε ήδη την ε, ε, διαπραγμάτευση και την εφαρμογή της Συμφωνίας Ναύτα για 20 χρόνια. Ε, νομίζω λοιπόν πως καλό θα είναι να λαμβάνονται υπόψη τέτοιου είδου υφιστάμενε συμφωνίες. Επίσης θα ήθελα στη δική μας έκθεση να περιλαμβάνονται περισσότερα σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει διεξοδική εξέταση αυτού του ζητήματος και θα πρέπει μεταξύ άλλων να αναφέρεται ότι χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα εφαρμόζει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά την συστηματική αξιολόγηση αυτών των ετών σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει στο μέλλον. Δηλαδή και σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όσο και σε ό,τι αφορά το κοινωνικό τομέα, αλλά και την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. το λόγο παρουσίασε διάφορες απόψεις. Επιτρέψτε μου να εστιάσω σε ένα θέμα. Είναι σημαντικό να μας απασχολήσει η ψηφιοποίηση των μελλοντικών συμφωνιών. Θα πρέπει να τη δούμε στο σύνολό της καθώς και τις αλλαγές που επέρχονται, θύματα, θέματα όπως ε, οι δύναμη της ψηφιοποίηση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα περισσότερο συνεκτικό τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια φιλελεύθερη ατζέντα με βάση κοινέ αξίες. Είπατε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε ένα διαφανή διάλογο με τους πολίτες μας και τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε μια ψηφιακή εποχή. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Είστε διευθύντρια του κλάδου εμπορίου. Ακούσατε πολλά. Thanks a lot, uh, Chairman Lange. Uh, thanks a lot. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα σχόλιά τους. Τα ακούσα όλα πάρα πολύ προσεκτικά, όλες τις παρατηρήσεις που διατυπώσατε και μια-δυο παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τα θέματα που θίξατε. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον εισηγητή και τον κύριο Τσαΐφη για τα σχόλια. Θα ήθελα καταρχάς να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο εκθέσεις. Ξέρετε ότι ως μέρος του πακέτου εμπορίου και όπως είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος Γιούνκερ, ετοιμάσαμε την ενδιάμεση έκθεση για όλες τις στρατηγικές. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική παραμένει αλλά κάνει μια αναφορά και σε θέματα που έχουν ήδη επιτευχθεί. Αλλά βεβαίως πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Πρόσφατα, και θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες ε, τις ε, ε, παρατηρήσεις ε, για την ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στην Επιτροπή και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής υπέβαλε την έκθεσή του για το θέμα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι βασικές αρχές της στρατηγικής παραμένουν προσπαθούν Ευχαριστούμε για ανοιχτού κανόνες που βρίσκονται στην βάση της ευημερίας μας που συλλαμβάνουν υπόψη τους το θέμα της κοινωνικής ε, προστασίας για να προωθηθούν οι ευρωπαϊκές αξίες. Όλα αυτά αποτελούν μέρος ε, της πολιτικής εμπορίου. Τώρα, το θέμα της ε, διαφάνειας, ένα θέμα που δείξατε αρκετή. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό σε ό,τι αφορά την νομιμότητα της εμπορικής πολιτικής. Ε, σημειώσατε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που δημοσιεύτηκαν τα σχέδια των εντολών από τις διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία το Σεπτέμβριο και για να επιτρέψουμε να διεξαχθεί συζήτηση στις χώρες μέλη με τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια αλλά και με τους πολίτες της χώρες μέλη. Δίχως άλλο, όλοι μας συνεχίζουμε να θέτουμε το ερώτημα στις χώρες μέλη να εμπλέξουν τα εθνικά κοινοβούλια σε θέματα πολιτικής. Επίσης ε, λέμε να ε, δημοσιευτούν τα παλιότερα, παλιότερες εντολές. Τώρα το δίκαιο εμπόριο για όλους. Εμείς απαιτούμε αμοιβαιότητα και ε, εξισορροπημένο εμπόριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και τις ε, συμφωνίες, όλοι ε, έκαναν παρατηρήσεις σχετικά με το, την πλευρά των εφαρμογών. Θα ήθελα να τονίσω ένα ή δύο σημεία. Καταρχάς, αυτή είναι η πρώτη έκθεση. Και δίχως άλλο θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αυτή είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι ιδανικά τα πράγματα του χρόνου θα μπορέσουμε να μάθουμε από τις εμπειρίες μας και να υιοθετήσουμε και τις παρατηρήσεις που έχετε την καλοσύνη να κάνετε. Προσπαθούμε να υιοθετήσουμε μια εξισορροπημένη στάση δεν θέλουμε να εικόνα που θα δημιουργήσουμε να είναι ρόδινη. Έχουμε παραθέσει καλά παραδείγματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομεί που βρισκόμαστε πίσω. Για παράδειγμα, η κρίση των ε, εμπορικών προτιμήσεων από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένους λόγους κατά την άποψή μας. Καταρχάς ε, δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση, υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης από πλευράς των επιχειρήσεων και αυτό ενθαρρύνει τα, ε, και εμείς ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να το κάνουν έχουμε και μία εντολή ως προς την παροχή περισσότερων πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας με βάση μία συγκεκριμένη σελίδα που συμβουλεύονται τα μέλη μας. Υπάρχουν πολύπλοκοι κανόνες που αφορούν την προέλευση και τώρα υπάρχει ένα ειδικό τμήμα και σε ό,τι φορά τη Συμφωνία ΣΥΤΑ υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν. Καταρχάς για να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να εξηγήσουμε στις εταιρείε πώς μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Τώρα, όπως μπορείτε να δείτε σε διάφορες χώρες μέλη, το επίπεδο χρήσης των προτιμήσεων διαφέρει. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε ε, τα διάφορα μέσα και η Επιτροπή με τις άλλες χώρες μέρη προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή των κρατών μελών σε αυτό το, ε, σε αυτό το θέμα. Α, τελείωσε ο χρόνος που είχα στη διάθεσή μου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σαϊφή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων που έλαβαν το λόγο και βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημείωσα τις παρατηρήσεις, αλλά πρέπει να διαπιστώσω ότι συμφωνούμε με πολλά σημεία που μας είναι σε όλους ιδιαίτερα σημαντικά, όπως παραδείγματο χάρη την εφαρμογή και την παρακολούθηση, την ε, ψηφιακές ε, εμπορικές συναλλαγές, την διαφάνεια, τις μιμιέ, τις οποίες πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα, τις ε, διάφορες επιχειρήσεις ε, και τους ε, ε, εργαζόμενους και όλο το άτομα που πρέπει να υποφελούνται από αυτήν την πολιτική. Πολύ πρακτικά όλα αυτά. Εγώ θα συνεχίσω στην εκπόνηση της εκθεσής μου. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για να λάβω υπόψη και περαιτέρω παρατηρήσεις και σχόλια πριν να ξαναπαρουσιάσω την εκθεσή μου στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η έκθεση θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο στις 22 Ιανουαρίου, φαντάζομαι λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι ολοκληρώσαμε και τη συζήτηση του σημείου 9 και περνάμε αμέσως στο 10. Πρόκειται για μια πολύ σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνόδου Κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Παναθηνικού Συνοβουλίου 27 και 28 Νοεμβρίου στο Αμπιτζάν, στην Côte d'Ivoire, στην αξία του Ελεφαντοστού. Θα μας ενημερώσει για την έκθεση αυτή η συνάδελφος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως ήμουν μέλος ε, εκ μέρου τη Επιτροπή μα στην Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Στιάνδη. Πρέπει να πω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μια συνάντηση που είχαμε δύο μέρες πριν από την διακυβερνητική αυτή σύνοδο κυβερνητική, ε, κορυφής. Οι συζητήσεις μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ήταν πολλά υποσχόμενοι, διότι υπάρχει κατά την άποψή μου καλύτερη προοπτική εκ των υστέρων να βρούμε κοινό έδαφος συνεννόησης μεταξύ ημών και ημών όταν συζητούμε. Και υιοθετήσαμε και ένα σύντομο μήνυμα για, προς την Σύνοδο Κορυφής λέγεται η έκκληση του Αμπιτζάμ και αφορά θέματα εμπορικά αλλά έχει και ένα ειδικό σημείο για τις επενδύσεις και το εμπόριο. Αναφέρεται στο μήνυμα αυτό ότι η ένταξη των αφρικανικών χωρών στα πλαίσια του, του ε, παγκοσμίου εμπορίου είναι προτεραιότητα και γι' αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί και σημασία μια υπηρετική εμπορική συμφωνία βάσει της συνεργασίας στις εμπορικές σχέση μεταξύ των χωρών. Είπαμε ότι μέσω της εμπορικής της πολιτικής θα πρέπει να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υλοποίηση αυτού του στόχου και οι αφρικανικές χώρες θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν σε θέματα προστασίας ε, το, της ε, προέλευσης κάποιων προϊόντων και άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν στα πλαίσια των ε, οικονομικών συνεργασιών βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, πράγμα που δεν είναι πάντα προφανές. Επίσης, οι αφρικανικές χώρες είπαμε ότι θα πρέπει να εγγυώνται και την νομική υπόσταση και νομιμότητα των επενδύσεων. Αυτό είναι και θέμα καλής διακυβέρνησης. Πολύ βουλευτές φαίνεται ότι συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν για την υπονάπτυξη τους και για την φτώχεια τους να ρίχνουν το βάρος σε όλους τους άλλους. Πρέπει και εκεί να υπομισθούν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν σε θέματα σωστής ε, διακυβέρνησης που είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει μια εποφελής εμπορική ε, σχέση και για τον αφρικανικό λαό γενικότερα. Αναγνωρίστηκε επίσης από την αντιπροσωπεία μας ότι το περίφημο σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων δεν είναι κάτι που αναφέρθηκε από τους ε, ε κοινοβουλευτικούς ε, ε, εκπροσώπους ούτε από τις κυβερνήσεις. Τα, 20, τα 55 περίπου κράτη που συμμετείχαν handled by Δεν γνωρίζουν ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μια ομάδα που αναπτύσσεται προοδευτικά. Έγιναν επίσης ε, διάφορες συζητήσεις και διαφορετικά αντιφατικά σημεία παρουσιάστηκαν ε, και από την κυρία Μογκερίνη για την ε, κοινωνία των πολιτών, για το ότι πρέπει να είναι παρόντες ε, οι εκπρόσωποι, ότι θα πρέπει να καλούνται να παρουσιάζουν και εκείνοι ένα μήνυμα την απόψη του τέτοιου είδου συνόδου κορυφή. Και είπαν ότι θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών των Αφρικανικών ε, κρατών να, είναι, να συμμετέχει περισσότερο. Αυτό είναι και ένα κριτήριο αξιοπιστίας των κυβερνήσεων. Τώρα, η δημιουργία θέσεων απασχόληση για του νέου Αφρικανού βεβαίω ήταν στον πυρήνα όλων των συζητήσεων. Δεν είναι εύκολη πρόκληση, διότι η αντιπροσωπεία μα πήγε στην ακτή του, ε, στο Ελεφαντόδοντο, στο Αμπιτζάν, στο ε, σχετικό γραφείο Εργασία για τους νέους και συζήτησε με πολλούς νέους Αφρικανούς οι οποίοι είχαν ε, ε, επαναπροωθηθεί από την Λιβύη στη χώρα τους. Οι περισσότεροι από τους νέους με τους οποίους μίλησα είχαν κάποιο επάγγελμα, ε, είχαν σπουδές, κατάρτιση, αλλά ήταν απολύτως σίγουροι ότι δεν θα ήταν σε θέση να, δουν, να βρουν στη χώρα τους ε, δουλειά. Και αν είχαν φίλους ή συγγενείς στην Ευρώπη, προσπαθούσαν όλοι να φτάσουν εδώ. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Ανάπτυξης γίνεται λόγος για, από τον Ειδικό Σύμβουλο για την Ανάπτυξη. Μιλήσαμε για τη Λιβερία, για τα ε, για την Λιβύη, όχι τη Λιβερία, διορθώνει ομιλήτρια. Ε, ξέρουμε ότι συμβαίνουν ακόμη ε, τρομερά πράγματα. Υπάρχουν τρομερές φωτογραφίες του τρόπου με τον οποίο κρατούνται κάποια άτομα. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν αυτή μια καλή βάση και προσέγγιση να συνεχίσουμε τις εμπορικές σχέσεις. Πρόεδρε, ίσως θα σε ευχαριστήσει να ακούσετε ότι πήγαν στην ίδια φυτεία μπανάνας και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ανάπτυξη, εκεί που πήγαμε και εμείς και η κυρία Ρενά. Και πραγματικά είδαν ότι υπάρχουν σοβαρές επιχειρήσεις που προφαρούν να κάνουν τη δουλειά τους με τρόπο που να είναι επωφελής και για τους λαούς που εκπροσωπούν. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση, Χάιντι. για την Τελωνιακή Ένωση των Αφρικανικών χωρών. Συζητήθηκε το θέμα αυτό. Ναι. Όχι στην Κοινοβουλευτική Σύνοδο Κορυφής. Έχω την εντύπωση ότι τα ε, κοινοβούλια είναι πολύ μακριά από την ε, εξουσία λήψης αποφάσεων. Οι κυβερνήσεις πιστεύουν ότι τα κοινοβούλια είναι κάποιες ε, οντότητες ε, μακρινές, εκτός της δικής τους δικαιοδίας. Εάν είχαμε το τελικό έγγραφο της Συνόδου ε, Κορυφής, ε, τα πρακτικά δηλαδή και τα αποτελέσματα, θα μπορούσα να σας δώσω κάποιες απαντήσεις, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμα. Μας είπαν από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Συμβουλίου ότι υπάρχουν ακόμη κάποια αμφιλεγόμενα θέματα ή κάποια τεχνικά θέματα και δεν έχει ε, συνταχθεί η έκθεση. Δεν μπορώ λοιπόν να σας δώσω απάντηση, αλλά πιστεύουμε ότι προχωρά αυτή η ε, συμφωνία όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ. Ωραία. Το έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να το συμβουλευτείτε ακόμα και στην περίπτωση αυτή κινούμεθα με πολύ γοργότερου ρυθμού από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τελειώσαμε λοιπόν με το σημείο 10. Περνάμε τώρα στο σημείο 11. Η συνεδρίαση του Διεθνούς ε, ε, Οργανισμού Εμπορίου θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο σημεία εισαγωγικά και μετά με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Επιτροπής. Καταρχάς, διεξάγεται μία συζήτηση για την Βίζα και πολλέ ΜΚΟ και δημοσιογράφους. Η έκθεση Εγκοστίνη απέριψε το 70% ε, τις ε, θεωρήσεις ε, και τη δυνατότητα να έχει κανείς πρόσβαση στο συνέδριο. Ήταν δύσκολο, δηλαδή να μπορέσει κανείς να παραστεί στη συνάντηση αυτή στο Μαϊρόμπι. Για μένα δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το συζητήσαμε και προηγουμένως ότι η εμπορική πολιτική απαιτεί διαφάνεια, απαιτεί διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Και θα καλούσα την Επιτροπή να πει ένα-δύο πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα. Εγώ έστειλα ως πρόεδρος μία επιστολή και είπα ότι κατά την άποψή μου όλα αυτά είναι αρκετά προσβλητικά. Τώρα δεύτερον, κοιτάζοντας σαν το ποντίκι, το φίδι, στρέφουμε το βλέμμα προς τις Ηνωμένε Πολιτείε και βλέπουμε τι κάνουν. Πήγανε δήλωση για, στις 24 Οκτωβρίου που με έναν ε, ε ε, άκομψο τρόπο είπαν ότι δεν θα πραγματευτούν πολλά από τα θέματα επιτάπητος ε, είναι στη διάθεσή μας για να συζητήσουν αλλά όχι για να διαπραγματευτούν. Ε, στο Μαρακέ σταμάτησε η προετοιμασία προκειμένου να υπάρξει ένα έγγραφο στη Γενέβη και νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε τι είναι αυτό το πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό για το πιθανό αποτέλεσμα που θα έχουμε στον Buenos Aires. Πηγαίνουμε εκεί με μια αντιπροσωπεία, ισχυρή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γίνει μια κοινοβουλευτική συνδιάσκεψη που ξεκινάει στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, αλλά από ό,τι φαίνεται όλα είναι υπό τη σκιά αυτού του ερωτήματος. Πώς μπορούμε να έχουμε την εγγύηση ότι θα επιτευχθεί κάποια πρόοδος, ότι θα υπάρξουν και νέα θέματα στην ημερησία διάταξη. Και αυτό σε ό,τι αφορά τις 164 χώρες ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού. Ο κ. Διντόνετ, διευθυντής της Επιτροπής και υπεύθυνο για το Διεθνές, ε, Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου, παρακαλείται τώρα να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι μια ενημέρωση θα σας ε, δώσω. Ε, δεν ξέρω από εκεί και μετά αν μπορώ να σας δώσω όλες τις απαντήσεις, αλλά θα είμαστε σε θέση με την επιτόπια, ε, αντιπροσωπεία μας εκεί. Ε, καθώς συζητήσατε αυτό το ζήτημα στην Ολομέλεια πριν από δύο εβδομάδες, θα ήθελα να σας δώσω όλες τις νέες πληροφορίες που έχουμε στο πλαίσιο της προπαραστευαστικής διαδικασίας, η οποία τρέχει κατά τι τελευταίες δύο εβδομάδες στη Γενέβη και έχει εντατικοποιηθεί. Έχουν υποβληθεί κάποιες νέε προτάσει από χώρε μέλη του ΠΟΕ. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση, ή περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με ε, πριν από δύο εβδομάδες σε ό,τι αφορά το αν θα καταφέρουμε τελικά να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης. Η θέση των κυρίων χωρών μελών ε, πράγματι οι θέσεις τους παραμένουν ε, διστάμενες. Δηλαδή και ακριβώς το γεγονό ότι εξακολουθούν να διείστανται απόψει τους θα καταστήσει δύσκολο το να φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τώρα στην υποστηρική διάσκεψη. Αλλά επιτρέψτε μου να σας αναφερθώ στα κυριότερα ζητήματα υποδιαπραγμάτευση των Buenos Aires και να σας πω ποια είναι η δική μα αίσθηση ως προς το προ τα πού θα κινηθούν διαπραγματεύσει στο πλαίσιο δηλαδή τη συνομιλία. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ενισχύσεων ε, ή επιδοτήσεων στον χώρο τη αλληλεία, ε, πράγμα ε, δηλαδή που αφορά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ η συζήτηση είναι πολύ ζωντανή και συνεχίζεται και σήμερα και αύριο θα συνεχιστεί στη Γενέβη. Εδώ λοιπόν θα μπορούσε ενδεχομένω να επιτευχθεί μια πρόοδο, ένα αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους κλάδους ή συγκεκριμένα είδη αφορα συγκεκριμένου κλαδου η συγκεκριμενα ειδη επιδοτησεων ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αλία IUU, αυτή την ε, λαθρέα παρανομική αναρχιαλία, και σε σχέση και με την εμπεραλίαυση των αποθεμάτων. Και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να προβούμε στη διαπραγμάτευση περαιτέρω ζητημάτων, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα ε, περιεκτικό αποτέλεσμα σε σχέση με αυτόν τον τομέα. Από εκεί και μετά υπάρχουν άλλε διαπραγματεύσει ό,τι αφορά γενικότερα τον τομέα τη γεωργία και εδώ συμμετέχουμε πολύ ενεργά από την πλευρά τη Ένωση, όπω είχαμε κάνει και στο πλαίσιο τη προετοιμασία για την 11η Υπουργική Διάσκεψη. Ε, και ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα είναι ε, η ε, δημόσια ε, συμμετοχή ε, στα κεφάλαια των αγροτικών επιχειρήσεων, δηλαδή το δημόσιο μέτοχος και εδώ τίθονται ερωτήματα μονίμων λύσεων, δικλείδων ασφαλείας, διαφάνεια σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και για μας το επίπεδο της φιλοδοξίας σε αυτό το τομέα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πακέτο, αν θέλετε, της συνολικής συμφωνίας που θα προκύψει από αυτή την υπουργική διάσκεψη. Ε, ειδικότερα στον τομέα της ε, γεωργίας, ε, το ζήτημα που έχει δημιουργήσει κάποιες εντάσεις είναι η δημόσια ενίσχυση υποστήριξη. Δηλαδή εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχει σύγκληση απόψεων και οπότε <clears throat> δεν είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει πρόοδος. Πέραν αυτών των δύο τομέων, όπου υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσει και αυτή την περίοδο, και έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδε, θεωρούμε πως ακόμα κι αν καταφέρουμε να καταλήξουμε σχέση με αυτά τα δύο σημεία, ε, δεν θα πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να ε, στοχεύσουμε προ μια συμφωνία, η οποία για παράδειγμα θα καλύπτει και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εδώ για παράδειγμα έχουμε προτείνει τη σύσταση μια νέα ομάδα εργασία ε, του ΠΟΕ, έτσι ώστε τα, οι χώρε μέλη να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται. Ζητήματα πάντοτε τα οποία αφορούν ακριβώ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου το πολυμερέ σύστημα εμπορίας και από εκεί και μετά ε, τα ε, ζητήματα ε, της, των υπηρεσιών και των σχετικών χώριων κανόνων σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και από εκεί και μετά το, τα ζητήματα διαφάνειας στο πλήρη των υπολογικών συναλλαγών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, θα υπάρξει μια συζήτηση σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την ανάπτυξη και την ε, περαιτέρω τον εντοπισμό των ζητημάτων που αφορούν το εμπόριο και την ανάπτυξη. Εμεί θα συμμετάσχουμε επικοδομητικά στη σχετική συζήτηση και θα υπογραμμίσουμε την ανάγκη εξατομικευμένων προσεγγίσεων σε αυτόν τον τομέα που θα βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά δηλαδή την διακριτική μεταχείριση ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των αναπτυσσόμενων χώρων. Πρόεδρε, αναφερθήκατε στο ζήτημα ε, το, του ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ζητήματα διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του ΠΟΕ, αλλά και με ζητήματα του μηχανισμού επίλυση διαφορών εκεί. Ε, και νομίζω πω είναι σαφέ πω σε ό,τι αφορά το ζήτημα του μη διορισμού μελών στο δευτεροβάθμιο ε, ε, όργανο, δηλαδή στο Appellate Body, θα αποτελέσει σίγουρα αντικείμενο ε, συνομιλιών των Υπουργών στο πλαίσιο της διάσκεψης. Και όπως είπατε και εσείς αλλά και η Επίτροπος Μάλστρομ στο παρελθόν σε σχέση με αυτό το ζήτημα, το εν λόγω θέμα δημιουργεί σοβαρή ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν δυνατό, θα μπορούσε δηλαδή να συμβεί, ε, ε, η, ε, πρόεδρος εκεί, η κυρία Μαρκόρα, ενδεχομένω να ε, ε, θελήσει να ξεκινήσει μια γενικότερη συζήτηση σε ό,τι αφορά τον μελλοντικό ρόλο του ΠΟΕ, ακριβώς όχι μόνο ως διαπραγματευτικό όργανο, αλλά και ως ένα όργανο διαβούλευσης, το οποίο θα μπορεί, μπορεί να λαμβάνει υπόψη του νέα ζητήματα, νέα θεματολόγια, ε, πράγμα βέβαια στο οποίο θα συμμετάσχουμε και εμείς ενεργά από την πλευρά της Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, γνωρίζουμε πώς θα διαρθρωθεί η συζήτηση, δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής του ΟΠΟ, ο κύριος Ρομπέρτο Αζεβέντο ανέφερε ότι θα υπάρξουν πέντε θεματικές συζητήσεις των Υπουργών ε, την πρώτη μέρα όπου θα καλυφθούν επιμέρους ζητήματα, ακριβώς η γεωργία, η ανάπτυξη, η θέσπιση κανόνων, ε, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλείας, ηλεκτρονικό εμπόριο και από εκεί και μετά μια σειρά από σε σχέση με τις υπηρεσίες και τη διαφάνεια. Από εκεί και μετά θα, υπάρχουν, θα αναλάβουν τον ρόλο των συντονιστών αυτών συζητήσεων επιμέρους υπουργοί και από εκεί και μετά ε, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της πρώτης ημέρα, θα υπάρξει μια ε, συζήτηση των δικών μας αντιπροσωπιών ε, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της συζήτησης της πρώτης ημέρας. Και από εκεί και μετά βέβαια το ποια θα είναι τα αποτελέσματα θα τα δούμε όπω όπως θα εξελίσσεται και πώς θα εξετάζεται η μερίσια διάταξη της διαστέψης. Τέλος, Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην απόφαση της κυβέρνησης της Αργεντινής να ακυρώσει ε, την πιστοποίηση των ε, ορισμένων μελών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ο Επίτροπος ε, ανέφερε και το κατέστησε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η εμπορική πολιτική να χαράσεται με έναν διαφανή αλλά και χωρίς αποκλεισμό τρόπο Κατά συνέπεια λοιπόν είναι σημαντικό η Υπουργική Διάστευση να βρίσκεται σε ε, διαλλαγή, να ακούσει τις φωνές από τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Προφανώς ε, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει η διάστευση να λάβει χώρα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και εμείς από την δική μας πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε και μέλη εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών μεταξύ μας. Ε, οπότε να πούμε ότι εμείς συμμεριζόμαστε τη δική σας άποψη αλλά και αυτή της Επιτροπής Προφανώ. και έχουμε ήδη κοινοποιήσει αυτή την τοποθέτησή μα ε, στην ε, κυβέρνηση τη Αργεντινή την περασμένη εβδομάδα, όταν τέθηκε δηλαδή αυτό το ζήτημα προ συζήτηση. Ζητήσαμε δηλαδή περαιτέρω εξηγήσει σε σχέση με αυτέ τι αποφάσει που έλαβε και το σκεπτικό που ακολούθησε και ακούσαμε ότι η Αργεντινή είναι διατεθειμένη να επανεξετάσει επιμέρου περιπτώσει εφόσον υπάρξει επικοινωνία των ε, σχετικών ε, ε, Υπουργείων από τις χώρες στις οποίες έχουν την έδρα τους αυτές οι ε, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Έκτοτε, εμείς λοιπόν έχουμε ενθαρρύνει ακριβώς τις ε, σχετικές ε, χώρε και οργανώσεις να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτές λοιπόν είναι οι κίνησει τις οποίες προβήκαμε και ε, να πούμε ότι εμεί από την πλευρά τη Επιτροπή έχουμε συνεχίσει να δίνουμε τι οδηγίε μα ε, τόσο στην ε, αντιπροσωπεία στη Γενέβη όσο και στην αντιπροσωπεία μα που βρίσκεται ήδη στον Πουένο Άρη για να λάβουν υπόψη τους αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ένα απλό ερώτημα. Επειδή ο κύριος Λάσερ δεν συμμετείχε στην προπαρασκευαστική συνάντηση στο Μαρακές και την κύρωσε την τελευταία στιγμή. Τι πιστεύετε εσείς θα έρθει τελικά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζουμε, ε, περιμένουμε ότι θα υπάρξει παρουσία σε υπουργικό επίπεδο. Θα υπάρξει διμερής δέσμευση και βεβαίως μια ευρύτερη δέσμευση αργότερα. Είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση να προωθήσουμε μερικά από τα θέματα και να αναζητήσουμε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης να δώσω το λόγο στον ε, Συμπρόεδρο. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί με αυτόν τον ε, νέο διαπραγματευτικό γύρο στον ΠΟΕ υπάρχουν και κάποιες ελπίδες οι οποίες δίνονται. Βέβαια, πολύ σωστά είπε ο πρόσωπος της Επιτροπής, ε, θα πρέπει να υπάρχει εδώ και μια πλατφόρμα για τις μικρο, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις έτσι ώστε να γίνουν ε, και οι δικές τους φωνές ε, αυτές και νομίζω πως είναι λυπηρό το γεγονό ότι δεν έχουν εμπλακεί στην όλη διαδικασία επαρκώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν ακριβώς τη βάση έτσι ώστε στο μέλλον να επιτύχουμε την δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας μελλοντικά στην Ευρώπη. Νομίζω πως είναι επίσης σημαντικό για μας να εξετάσουμε το πώς μπορεί να τεθεί επιτάπητος ε, το Doha Development Νομίζω πω δηλαδή σε σχέση με αυτόν τον ε, ε, γύρο θα πρέπει να θέσουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο τη συζήτηση. Στόχοι δηλαδή οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για εμά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο και του Ταμείου για την Αφρική και τα νέα εργαλεία χρηματοδότηση που έχουμε στη διάθεσή μα. Άρα λοιπόν το Ταμείο που έχουμε δημιουργήσει για την Αφρική θα πρέπει να ε, αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του νέου διαπραγματευτικού κύκλου, όπως κάναμε και στο πλαίσιο ε, του ΕΦΣΙ, δηλαδή του ε, Ταμείου για τις ε, διαθροτικέ επενδύσει. Ε, και από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά το στόχο, για παράδειγμα την πρόσβαση στην ίδρυυση και τα συστήματα αποχέτευση ή τον στόχο 7 σε σχέση με την ανανεώσιμη ενέργεια, δεν θα χρειαστούμε κάποια ε, γενικότερα πλαίσια τα οποία θα δημιουργήσουμε σε ό,τι αφορά την συνεργασία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτέ τι χώρε και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν πω τέτοιου είδου συνεργασίε, ειδικότερα στι υπαίθριε περιοχέ, θα μα έδιναν τη δυνατότητα να εμπλέξουμε όλους τους ε, ε, ε, ανθρώπους, ε, όλους τους πολίτες αυτών των χωρών αντί να χρειάζεται να μεταναστεύουν από την επαρχία στις ε, πόλεις να ζουν μέσα σε σλάμ, σε παρακουπόλεις και στη συνέχεια να βρίσκονται στα δίχτυα των δικτύων προώθησης της λαθρομετανάστευσης. Εκείνο που θα με ενδιαφέρει να ακούσω από την Επιτροπή είναι πώς προσπαθούμε να αναφερθούμε σε ζητήματα που μας απασχολούν στο πλαίσιο των ημερών συμφωνιών εμπορίου ε, σε αυτή τη συζήτηση ε, στον ΠΟΕ. Μήπως δηλαδή θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια βάση προσυζήτηση και στη Γενέβη. Ε, και νομίζω πως η δική μας αρμόδια υπηρεσία έχει συντάξει ε, μια σχετική ε, μελέτη ως προς το ποιες κατευθυντήρες γραμμές θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ακριβώς σε σχέση με τις σημερινές συμφωνίες που συνάπτουμε. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ότι στο πλαίσιο της, της διαπραγμάτευσης του Brexit βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Έγινε και μια κλεισμένο το θηρό ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας. Οπότε εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι, θα μας απασχολήσει το ζήτημα του Brexit στο Buenos Aires και πώς θα τοποθετηθεί σε σχέση με αυτό το ζήτημα η Επιτροπή. Ποια θα είναι η θέση που αθετήσει, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αν ερωτηθεί. Ευχαριστώ. Κυρία Ροντρίγκη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ και τον προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι πάντα είναι υπέρ ε, ε, των θεμάτων αυτών της ε, πλευρών ε, πολιτικών αυτός που ακολουθούμε και πάντα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να μου πείτε, σε σχέση με το διατητικό δικαστήριο και αυτό που σας απασχολεί σε σχέση με μας όσον αφορά τις κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί. Ποιες είναι οι προοδοκίες σας, πιστεύετε ότι θα μπορέσει να επιληθεί το θέμα, πότε και με ποιο τρόπο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαιτέρως η Επίτροπος κάνει μεγάλες προσπάθειες ώστε να γίνει, έχει αυτή πολύ πολύπλευρη διάσταση η οδηγία για το εμπόριο. Θα ήθελα να μου πείτε εάν στην διάσκεψη των Υπουργών αυτή θα προσπαθήσετε ε, σε σχέση με το θέμα αυτό να έχετε με το μέρος σας και περισσότερες χώρες. Και τελικά κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την ε, πολυμερή συμφωνία επενδύσεων, τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Ο Κλάους Μπούχνα έχει το λόγο. Ναι, θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν, Επιχαίρω το γεγονό ότι αναφέρθηκε το ζήτημα ε, τη ε, μη συμμετοχή, ε, εν πάση περιπτώσει τη δυνατότητα συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θεωρώ πω είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή του για την επιτυχή έκβαση αυτή τη διάσκεψη και θα πρέπει λοιπόν και είναι σημαντικό το ότι περιλαμβάνουμε στη δική μα αντιπροσωπεία εκπροσώπου από των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του διαπραγματευτικού γύρου τη Ντόχα, αναφέρθηκαν ήδη αυτά, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση της Επιτρόπου Μάλιστον. Δηλαδή, θα ε, φροντίσει έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια επιτυχία έκβαση σε ό,τι αφορά ε, την Τόχα. Γνωρίζετε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει, δεν θα τις επαναλάβω. Γνωρίζετε και ποια είναι η τοποθέτηση της ε, αμερικανικής πλευράς, οπότε θα ήθελα να ακούσω ποια θα είναι η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως θα εκπροσωπηθεί από την Επιτροπή Μάλιστον. Και τελευταίο ερώτημα από την πλευρά μου. Αναφέρθηκε τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από άλλε χώρες μέλη της, ε, του ΠΟΕ ότι θα ήταν καλό να συσταθεί μια ομάδα εργασία σε ό,τι αφορά το e-commerce, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά υπήρξαν πολύ ε, κατηγορηματικέ αντιδράσει από άλλε χώρε μέλη. Υπόθηκε δηλαδή ότι θα πρέπει ουσιαστικά ε, να επανέλθουμε στη φάση τη διαπραγμάτευση και τη συζήτηση που βρισκόμασταν το 1989. Οπότε ποια είναι η θέση τη Επιτροπής, πώς θα κινηθούμε σε σχέση με αυτό. Ε, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και ο Χέλμουντ Σόλς στο δεύτερο λόγο. Ευχαριστούμε για αυτές τις ε, Επιτρέψτε μου να θέσω σε δύο ακόμα ζητήματα ε, συμπληρωματικά προς αυτά που ανέφεραν συνάδελφοι και για τα οποία τους ευχαριστώ ειδικότερα σε ό,τι αφορά δηλαδή και τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και γενικότερα την εκπροσώπηση της κοινωνίας ε, των πολιτών. Ελπίζω δηλαδή από τεχνικής άποψης να καταστεί δυνατό τελικά να συμμετάσχουν όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι. Ελπίζω εδώ δηλαδή να αναθεωρήσει και η κυβέρνηση της Αργεντινής την άποψή τη μετά από τις πιέσεις που έχουν ασκηθεί. Πέραν λοιπόν όλων αυτών να πω ότι έχουμε συζητήσει τα διάφορα ζητήματα, τι διάφορες πτυχέ, για παράδειγμα την Τόχα, ε, τα νέα θέματα που έχουν τεθεί προς διαπραγμάτευση και ούτω καθεξή. Αλλά από εκεί και μετά, σε ποιο βαθμό και πόσο σοβαρά ε, λαμβάνει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή και την, ε, τις αντικές αντιδράσεις ε, άλλων χωρών μελών, ε, προκειμένου να επιτευχθεί τελικά μια συμφωνία. Δηλαδή πόσο είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει εδώ τον ηγετικό ρόλο για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Γιατί αν κανεί δεν τον αναλάβει θα είναι δύσκολο να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Εάν δηλαδή ο γύρο τη Ντόχα δεν ολοκληρωθεί επιτυχώ, ουσιαστικά θα υπονομευθεί το όλο σύστημα του Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πούν ότι εμεί μπλοκάρουμε, δεν επιθυμούμε, ενώ οι υπόλοιπε χώρε θα πούν ότι αν δεν υπάρξει ολοκλήρωση σε σχέση με την Τόχα, ούτε εμεί θα θέλουμε άλλη πρόοδο, θα μπλοκάρουμε κι εμεί. Άρα, τι κάνει η Επιτροπή έτσι ώστε να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή το χειρότερο σενάριο, αν θέλετε. Ε, δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω. Η θέσπιση κανόνων. Εμεί στην ε, Steering Committee, στην Επιτροπή δηλαδή Καθοδήγηση του ΠΟΕ, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα την ανάγκη της, ε, ενός αυξημένου ε, κοινοβουλευτικού χαρακτήρα του ΠΟΕ, δηλαδή περισσότερη σύνδεση με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών που συμμετέχουν στον ΠΟΕ. Νομίζω πως ε, σε ό,τι αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε σε καλή θέση, γιατί ακριβώς η κυρία Μάλστρομ έρχεται τακτικά στο κοινοβούλιο και μας ενημερώνει. Οπότε δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοχλό άσκηση πιέσεων αυτό ο αυξημένο κοινοβουλευτικό χαρακτήρας του ΠΟΕ στο μέλλον έτσι ώστε να αποφεύγουμε προβλήματα και να επιτύχουμε ένα ε, βήμα προς τα μπροστά στο μέλλον σε ό,τι αφορά την επίλυση δύσκολων ζητημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Και ε, για την προπαρασκευή τη της υπουργικής υπάρχει η σχετική συζήτηση ε, όπου οι διάφοροι συμμετέχοντες θα ε, εκφράσουν την άποψή τους. Οπότε ε, ποια θα είναι η άποψη της Επιτροπής, θα ταχθεί υπέρ αυτής της περισσότερης, του περισσότερου κοινωνικού, αν θέλετε, κοινοβουλευτικού χαρακτήρα του ΠΟΕΣ στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να δώσω τώρα και πάλι το λόγο στην Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πολλά, πολλά τα θέματα. Ενδεχομένως ε, θα μπορούσαν να απαντήσω σε μερικές από τις άμεστες ερωτήσεις που μας απευθύνεται. Να ξεκινήσω από το τέλος. Τώρα, το πώς προσεγγίσουμε το όλο θέμα της ε, εντολής και του γύρου της Ντόχα. Εμείς περιμένουμε ότι η Υπουργική Συνδιάσκεψη θα θέσει την ημερησία διάταξη για τα επόμενα δύο χρόνια. Και για μας είναι αυτός ο στόχος να επιτευχθεί. Για μας σημαίνει ότι θα συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις σε μία, ως προς μία σειρά από θέματα που έχουν σχέση με την δήλωση της ΔΟΧΑ. Δεν αλλάξαμε την άποψή μας από την δέκατη υπουργική ε, συνδιάσκεψη το, το Ναϊρόπι λέει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις εντολές διαπραγμάτευσης. Εμείς επιβεβαιώσαμε ότι θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε μερικά από αυτά τα θέματα και θα προσπαθήσουμε η πρόοδος μας να είναι ε, εκθετική. Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπόψη της και άλλα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Εδώ τίθεται και το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα θέλαμε στη συνδιάσκεψη να γίνει ένα βήμα μπροστά ως προς αυτό το θέμα. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα θέματα που θέσατε σαφώς είμαστε υπέρ της κοινοβουλευτικής διάστασης δηλαδή η διάσκεψη αυτή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των πραγμάτων μέσα στην οργάνωση αυτό απαιτεί γιατί εμείς να αρχίσουμε την, να διοχετεύσουμε την απαραίτητη ενέργεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι φορά τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για ένα θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί από τις διάφορες οπτικές γωνίες του ΠΟΕ. Ε, το ΠΟΕ έχει πολλές λειτουργίες ελέγχου, ε, διαχείρισης Όλες ε, λοιπόν αυτές οι αρμοδιότητες ε, χρειάζονται μία αναβάθμιση έτσι ώστε ο ΠΟΕ να μπορεί πιο εύκολα να συνάπτει συμφωνίες. Και μετά ξεκινάμε με μερικά βασικά θέματα. Διαφάνεια, αύξηση της διαφάνειας ε, στο σύστημα. Και εσείς υποβάλλατε μια πρόταση από αυτή την άποψη. Άλλοι, αναφερθήκατε στις Ηνωμένε Πολιτείε, αναφέρουν ότι προσπαθούν ε, να επιτύχουν καλύτερες μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι προτάσεις δεν έχουν ακόμα διατυπωθεί. Θα δούμε αν τα μέλη θα υποβάλουν συγκεκριμένες ε, προτάσεις για το ΠΟΕ. Και εμείς με τη σειρά μας θα μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε όλα αυτά όταν διατυπωθούν πλήρως. Δεν είναι απόλυτα σαφές πότε και πώς το ερώτημα των συναντήσεων με τον ανώτατο φορέα θα επιληθεί. Υπευλήθη μια πρόταση να προχωρήσει η διαδικασία για τις τρεις θέσεις που χειρεύουν. Αυτό όμως δεν υποστηρίχθηκε από συνένεση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ε, τη ρύθμιση διαφωνών. Για μας ε, αυτό είναι ένα θέμα μεγάλου προβληματισμού. Αν δεν ληφθεί κάποια δράση, το θέμα αυτό δεν θα λυθεί από μόνο του, το αντίθετο θα έλεγα. Θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο, θα γιγαντωθεί από τη στιγμή που θα προκύψουν ακόμα περισσότερες χειρεύουσες θέσεις. Στα πλαίσια της συνδιάσκεψης που είναι μια ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα να συγκεντρωθεί πέρα από το θέμα των διαπραγματεύσεων και την ημερησία διάταξη της ίδιας της διάσκεψης θα συναντηθούμε διμερώσει στα πλαίσια μικρών ομάδων και με άλλους εταίρους Θα μιλήσουμε για την Εθνική Πρωτοβουλία κατά των ε, βασανιστήριων. Εδώ μιλάμε ότι θα πρέπει να προωθηθούν τα προγράμματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία που θα πρέπει να διερευνήσουμε. Αυτές οι συζητήσεις έγιναν και ξεκίνησαν στα πλαίσια του Wincy Trial, της δίκης Wincy, UNC Trial θα συνεχίσει διερκής, ε, ε, θα συνεχιστεί το ενδιαφέρον ε, και μετά και πριν το MC11. Πιστεύω ότι απάντησα σε όλα τα σημεία. Ζητάω συγγνώμη αν κάποιο ξέχασα. Ευχαριστώ. Βεβαίως θα υπάρξουν πολλές διμερείς συνεδριάσεις και αυτή θα είναι μία από τις πιο σημαντικές. ένας Γερμανός καθηγητής κοινωνιολογίας, ο Σκανίκ, έγραψε ένα βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο Buenos Aires. <clears throat> Πολλοί από τους παριστάμενους θα είναι μέλη της αντιπροσωπείας. Καλό ταξίδι. Θα τα πούμε στο Buenos Aires στο 12 που είναι το αγαπημένο μου, είναι τα διάφορα. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι σε 10 λεπτά πάμε για ένα ποτό στο εστιατόριο Origin. Είναι στο κτίριο ε. Θα πρέπει να πάρετε το σανσέρ, να πάρετε το ε, να κατεβείτε στο Μεντάν και μετά ξαναπάτε το Σασένα, πάτε στον πρώτο όροφο. Ναι, ναι, είναι ένα ισπανικό εστιατόριο. Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται για τον Ιανουάριο. Ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε για τα Χριστούγεννα και τον καινούριο χρόνο.